Αγαπητοί συνάδελφοι. Προτείνω να ξεκινήσουμε. Θα έρχεται και ο Πρόεδρος, φαντάζομαι. Δεν ξέρω πού είναι ακριβώς. Μπήκα αμέριμνη στην ε, αίθουσα, θεωρώντας ότι θα περάσω μια ήρεμη πρωινή συνεδρίαση και ξαφνικά δάμε στην Προεδρία. Λοιπόν, έχουμε τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και την ανάκληση της αποφάσης πλαίσιο 2005-222 με την κυρία Χολμάιερ. Μέτρο το οποίο αφορά ουσιαστικά την εναρμόνιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Θα ακούσουμε την ενημέρωση από το Συμβούλιο και μετά από τον κύριο Ερνάντες Μπαταγέρ φανταζομαι ε, ότι προφέρω και σωστά το, το όνομά σας. Και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Αλλά πρώτα βέβαια την κυρία Χολμάιερ θα ακούσουμε παρακαλώ. Η συγγήτρια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα σας δώσω μια πολύ σύντομη ενημέρωση για τις εξελίξεις στην ε, υπόθεση αυτή. Έχουμε την έκθεση που ε, κατατάθηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο Εν τω μεταξύ, πραγματοποίησαμε αρκετέ και πολύ ενδιαφέρουσε συνεδριάσει και επαφέ ε, τόσο με του δικαιώδει ηγητέ όσο και με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να πω ότι κάποια σημεία τα συζητήσαμε πολύ εντατικά στι συναντήσει αυτέ. Θα σα τα αναφέρω εν συντομία καταρχά την διεύρυνση τη νομική βάση, το ενδεχόμενο δηλαδή, την ανάγκη να διευρυνθεί η νομική βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζήτησε ο κύριος Άλβαρο κυρίως, αλλά και ο κύριος Άλμπρεχτ θεωρώντας ότι η πρόληψη ως θέμα είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό τουλάχιστον μέσα στην οδηγία αυτή. Επίσης είχαμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αστυνομική, τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών. Είχαμε επίσης θέματα κυβερνοεπιθέσεων από κράτη εις βάρος κρατών Και κάτι άλλο το οποίο δεν συζητήθηκε ε, ρητά, αλλά φαίνεται ότι θα βγουν τα κράτη από το πεδίο εφαρμογής και ζητήματα πρόσβαση σε μία ασφαλή ε, δίκτυα ψηφοφόρων. Επίσης έχουμε ζητήματα επιθέσεων, ε, έκνομων επιθέσεων ε, σε δεδομένα Φερρυπίν ε, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. και ορισμούς του υλικού που θα περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής του ε, νέου κανονισμού. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί ορισμοί στα διάφορα κράτη-μέλη και έτσι τώρα μέσα στην οδηγία δεν είναι σαφές ακόμη ε, το τι ισχύει. Ένα άλλο θέμα που συστήσαμε ήταν οι ή λόγοι μετρίασης της ποινής ή οι επιβαρυντικές περιστάσεις και άλλα αντίστοιχα ζητήματα τα οποία λίγο πολύ πρέπει να διευκρινιστούν. Επίσης έχουμε και από άλλες επιτροπές αντίστοιχα παρακολούθηση της υπόθεσης. Εμείς έχουμε επίσης να πάρουμε τη γνωμοδότηση Επιτροπής Βιομηχανίας, Προϋπολογισμών Εξωτερικών κτλ και περιμένουμε να δούμε τις δικές τους θέσεις. Είναι πολλά τα προβλήματα. Επί παραδείγματι στη Γερμανία έχουμε ένα εκατομμύριο Τρόιανς, ε, δουριουσίπους δηλαδή το μήνα, σε επιθέσεις κατά του τραπεζικού συστήματος. Είναι πολλά, όπως είπα, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και και η αύξηση των επιθέσεων μέσω του ίντερνετ. εις βάρος των ε, οργανισμών μας, των φορέων μας ή των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ενδιαφέρον είναι δε ότι χώρες του, κόσμου όπως η Βραζιλία ε, δαπανούν πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς για την ασφάλεια του ε, ίντερνετ. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 25 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες ζημιά ε, το χρόνο από τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι, πολλές, είναι πολυδιάστατο λοιπόν το θέμα. Θα πρέπει να δούμε όλες αυτές τις πτυχές του. Και ευχαριστώ τόσο το Συμβούλιο όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ειλικρινή συζήτηση των ε, θεμάτων. Το cloud computing είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Αναφέρεται μέσα στην οδηγία και θεωρούμε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον εάν ε, πρόκειται να περάσει αυτή η οδηγία και να υλοποιηθεί, να περιλαμβάνει την τελευταία το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης τεχνολογίας, δηλαδή να έχει αρκετή κάλυψη και του cloud computing. Γι' αυτό λοιπόν Όπως είπα, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Είναι πολλοί ορισμοί, δεν έχουν κλείσει όλα τα θέματα ακόμα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η κυρία Γκάραε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της ε, Ουγγρικής Προεδρίας, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το στάδιο των αισιών στο Συμβούλιο. Είμαι πρόεδρος της ε, αντίστοιχης ομάδας εργασίας που εξετάζει το θέμα επί Ουγγρικής Προεδρίας. Η Προεδρία ε, έχει, είναι προσιλωμένη στους ε, στόχους της οδηγίας ε, στην καταπολέμηση δηλαδή του εγκλήματος του κυβερνοχώρου. Βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας το θέμα αυτό. Οπότε οργανώσαμε στη Βουδαπέστη στα μέσα Απριλίου μια υπουργική διάσκεψη υψηλού επίπεδου και παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά όλες τις εξελίξεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε πολύ ειλικρινείς στην ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης να σας καθησυχάσω το Συμβούλιο θεωρεί πάρα πολύ χρήσιμες αυτές τις ανταλλαγές, αυτό το διάλογο, συνεπώς θα ενημερώνεστε τακτικά και ειλικρινά και από τη δική μας πλευρά για να προετοιμάζετε καλά και τη δική σας θέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χολμάιερ, την εισηγήτρια που έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ζήτημα αυτό και έχει μεριμνήσει για την επιτυχία των προσπαθειών. Συνεπώς ε, ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουν συζητήσεις ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Ε, θα ήταν επιτυχία αν υιοθετούσαμε μια κοινή άποψη στις 10 Ιουνίου στο Σύμβουλο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Θέλουμε το θέμα αυτό να συζητηθεί στο Συμβούλιο του Ιουνίου και προσπαθούμε να ε, καθορίσουμε μια κοινή προσέγγιση σύμφωνη σε μεγάλο βαθμό με τα συμπεράσματα ε, του Απριλίου όπου έλαβε χώρα ένα ακόμα Συμβούλιο Υπουργών. Είχαμε τότε ετοιμάσει ένα έγγραφο για αυτό το Συμβούλιο και με βάση αυτό το έγγραφο θέλουμε ε, να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι έχετε πρόσβαση αυτό το έγγραφο, οπότε γνωρίζετε τις λεπτομέρειες και μπορείτε να διαπιστώσετε ε, ποια ήταν τα τελικά συμπεράσματα του Συμβουλίου αυτό το ζήτημα. Ε, νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο να το διαβάσετε. Να πω δύο λόγια και για το κείμενο το ίδιο. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το νομοθετικό κείμενο. Πρώτον, διότι χρειάζεται να προσαρμοστούμε στη Λισαβόνα. Υπάρχει μια απόφαση πλαίσιο που υιοθετήθηκε με συγκεκριμένους κανόνες. Αυτή η οδηγία τώρα θα ήταν ένα βήμα μπροστά, διότι θα επέτρεπε στην Κομισιόν και σε άλλους να διαπιστώσουν πώς προχωράει η εφαρμογή. Ταυτόχρονα μας επιτρέπει να στείλουμε και ένα πολιτικό μήνυμα. Τι είδους πολιτικό μήνυμα? θέλουμε να αυξήσουμε τις προσδοκίες των κρατών μελών και των πολιτών μας σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του κυβερνού εγκλήματος. Θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία κρίσιμων υποδομών. Αυτό προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις πολύ νωρίς ήδη. Ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία συμπεριλάβαμε στο προσχέδιο της δικής μας ε, πρώτας τροπολογίας. Η προστασία αυτών των υποδομών αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα επιθέσεις εναντίον ε, τραπεζών. Ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών. Είναι πολύ σημαντικό να τις πολεμήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε και τις επιθέσεις botnet, botnet ε, άρνησης εξυπηρέτησης. πιστεύουμε ότι και αυτές οι επιθέσεις αποτελούν ε, σημαντικό πρόβλημα και ε, είναι επιβαρυντικό στοιχείο. Ε, θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η οδηγία αυτή θα είναι οδηγία που θα εμπίπτει στο ποινικό δίκαιο. Συνεπώς θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις γνωρίζοντα το. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μιλάμε για μια οδηγία ποινικού δικαίου λοιπόν, το οποίο σημαίνει ότι διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. Θα πρέπει να υπάρχει μια νομική βάση κατάλληλη και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε 10 χρόνια ε, θα εξακολουθεί να εφίσταται. Γιατί αλλιώς ε, δεν θα είναι καλή νομοθετική τεχνική να την ε, δεχτούμε ως νομική βάση. Αυτά καλή επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στηριζόμαστε σε εσά, στη συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε. Thank you. thank Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Γιάκου Μπορατίνσκι από την Κομισιόν. Thank you very, much, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, μάλλον δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η Προεδρία ήταν πολύ ικανοποιημένη με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η διαδικασία των συζητήσεων της οδηγίας. Εκτιμήσαμε συνάντηση που είχαμε πρόσφατα με συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, του εισηγητού και των σκιωδών. Πολλά θέματα που ανέφερε και ο Χρυμάγερ συζητήθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό για μας η οδηγία που θα εγκριθεί τελικά να δίνει προστιθέμενη αξία εν συγκρίση με τα παρόντα. Η Προεδρία ανέφερε μια θετική τροποποίηση που έλαβε χώρα. Δεν έχουμε φτάσει στην τελική φάση των εργασιών του Συμβουλίου. Πιστεύουμε ότι ένα σημείο ενδεχομένω ίσως να μην συμπεριληφθεί. Το θέμα του spoofing. Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε περαιτέρω. Σωστά, τα μέλη του Κοινοβουλίου δεν υπερέβαλαν τις προσδοκίες όσον αφορά το εργαλείο αυτό του ποινικού τομέα όσον αφορά την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο. Το ποινικό αυτό εργαλείο είναι ένα από τα πολλά στοιχεία της εικόνας που από μέτρα πολιτικής που μπορούν τελικά τα μέσα αυτά να κάνουν τη διαφορά, αλλά οι προσδοκίες των ευρωβουλευτών που θέλουν να τονίσουν την καταπολέμηση των εγκλημάτων του κυβερνοχώρου και πρόληψη αυτού είναι θεμητές ανησυχίες στα πλαίσια της συζήτησης λοιπόν, το Κοινοβούλιο θα λαμβάνει γνώση, θα συζητούμε διάφορα μέτρα κατά πολεμήσεως εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, αυτό θέλαμε και γι' αυτό δώσαμε κάποια έγγραφα στην Γραμματεία, όπως στρατηγητή για την εσωτερική ασφάλεια, όπου τα εγκλήματα του κυβερνοχώρου είναι ένας από τους πέντε βασικούς στόχους. Προτεραιότητα για θέσπιση μέτρων και γενικότερα το, η ψηφιακή ατζέντα προχωρά πιο πέρα από το θέμα της ασφαλείας στο διαδίκτυο και μόνο. Δημιουργεί ένα πλαίσιο πολιτικής για την όλη συζήτηση. Όπως είπε η Προεδρία, υπάρχουν όρια όσον αφορά τα ποινικά μέσα, όμως είναι καλό ότι μπορούμε να συζητούμε αυτά τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί. Είτε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Εγκλήματα του Κυβερνοχώρου, είτε σειρά άλλων μέτρων που ευαισθητοποιούν τους πολίτες όσον αφορά τους κινδύνους του διαδικτύου. Τώρα είναι κάτι πέρα από τη δική μου Γενική Διεύθυνση των Εσωτερικών. Ε, ίσως μπορούν να συζητηθούν και οι θετικές υποχρεώσεις της βιομηχανίας πληροφορικής. Δηλαδή να συμπεριλαμβάνει είτε σε λογισμικό είτε σε εξοπλισμό υλικό μέτρα ασφαλείας. Ούτω ώστε να είναι πιο ασφαλής η δραστηριότητα των πολιτών όταν σε το διαδίκτυο online. Είναι θέματα προς συζήτηση. Περιμένουμε αυτή τη συζήτηση κατανοώντας ότι σε αυτό, με αυτό το μέσο για ποινικά μέτρα ίσως δεν μπορούμε να επεκταθούμε επαρκώς όσον αφορά το ζήτημα της πρόληψης σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω τη συζήτηση με την... ΕΕ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κύριος Ερνάντες Μπαταγιέρ και μετά μπορούμε να δώσουμε το λόγο στα μέλη, τους ευρωβουλευτές που θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Κύριε gracias. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση και εκ μέρους του ΕΜΟΥ του ίδιου βέβαια, αλλά και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να παραστούμε και να σας παρουσιάσουμε την έκθεση που υιοθετήσαμε στις 4 Μαΐου. Και αφορά αυτήν ακριβώς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν, συμμεριζόμαστε την ανησυχία της Κομισιόν για το μέγεθος και το εύρος της ε, απειλής, καθώς ε, επίσης και την ανησυχία για τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει και τις ζημίες αυτή η απειλή. Οπότε δεχόμαστε, υποδεχόμαστε θετικά την πρόταση οδηγίας και τα πρόσθετα μέτρα, μη νομοθετικά μέτρα, τα οποία αφορούν μια συντονισμένη δράση και την πιο αποτελεσματική εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την πρόταση οδηγίας, πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η επικαιροποίηση των ορισμών ε, των αδικημάτων, επίθεση εναντίον συστημάτων πληροφορικής, καθώς επίσης είναι σημαντική και η βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να διευρύνουμε αυτό το συντονισμό τόσο στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όσο και σε ορισμένα στοιχεία τα οποία καλύπτει ο συντονισμός. Θεωρούμε ότι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη είναι απόλυτα σημαντική για την ψηφιακή οικονομία. Το κόστος, το ετήσιο κόστος αυτή τη στιγμή των κυβερνών εγκλημάτων είναι τεράστιο. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η οδηγία να αντικατοπτρίζει την σοβαρότητα αυτών των αδικημάτων και να δίνει ένα αποτρεπτικό μήνυμα προς αυτούς έναν των οποίων οι πολίτες μας ζητούν αυξημένες εγγύσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια κλιμάκωση των ποινών σύμφωνα σε συνάρτηση με την σοβαρότητα του αδικήματος. Είναι η αρχή της αναλογικότητας των ποινών, των κυρώσεων, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτριστεί και στην οδηγία. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των αδικημάτων, θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικό, τέρος, το αδίκημα ε, ε, της ε, ε, παράνομης παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών. Θέλουμε να καλύπτονται επίσης οι επιθέσεις μέσω δικτύων ζόμπι, καθώς επίσης και τις επιθέσεις DNS ε, και να καλύπτω και επιθέσεις DNS, δηλαδή ε, άρνησης εξυπηρέτησης. Η Κομισιόν μέχρι τώρα λέει ότι μόνο 17 από τα 27 κρατη έχουν επικυρώσει το, τη σύμβαση της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον χώρο. Ζητούμε και από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση το συντομότερο δυνατό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε την νομική βάση για όλη την Ευρώπη. Αναγνωρίζουμε ότι είναι επίγουσα αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά θα επιθυμούσαμε η Κομισιόν να ε, ετοιμάσει μια συνολική προσέγγιση για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Να μην περιορίζεται δηλαδή μόνο στην τιμωρία, αλλά θα πρέπει στην πρότασή της να συμπεριλάβει και την πρόληψη και την κατάρτιση και ενημέρωση. Λαμβάνοντα υπόψη και την στρατηγική της Ευρώπης 2020 και την ψηφιακή ατζέντα. Υποστηρίζουμε όλα τα προγράμματα κατάρτισης και τις συστάσεις καλών πρακτικών που προτείνονται για να ενισχυθεί το δίκτυο των σημείων επαφής που υφίσταται 24 ώρες το 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Προκειμένου να ενισχύσουμε επίσης την άμυνα της Ευρώπης έναντι των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ε, μια ένωση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία θα ενταχθούν οι εργασίες της ΕΝΙΣΑ και της ΣΕΡΤ. Επίσης, θα πρέπει να επιμείνουμε στην πρόληψη με πιο κατάλληλα μέτρα. Οι κατασκευαστές εξοπλισμού θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες έτσι ώστε τα προϊόντα τους να είναι πιο ασφαλή. Θα πρέπει να εξετάσουμε δηλαδή τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτότητας για όλη την Ευρώπη. Καλοσχεδιασμένο βέβαια, προκειμένου να αποφύγουμε ε, τις παραβιάσεις της προσωπικής ζωής. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις ικανότητες του IPUV6 και την κατάρτιση στην προσωπική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, που θα έπρεπε να είναι ένα σημαντικό κομμάτι οποιοδήποτε, οποιασδήποτε μελέτης για, την για τον ψηφιακό αλφαβητισμό θα πρέπει να ενισχύσουμε ένα ευρωπαϊκό τομέα ασφάλειας των πληροφοριών που θα πρέπει να είναι ισχυρός, ικανός, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί με τον αντίστοιχο των ΗΠΑ που χρηματοδοτείται πολύ. Τέλος, θα πρέπει να αυξήσουμε σημαντικά τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς επίσης και κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Θα πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση να χρηματοδοτήσουμε έρευνα και ανάπτυξη για την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και απόκρισης για την απάντηση σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Τέλος, θεωρούμε ότι οι τελευταίες ε, τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα πληροφορικής και ε, αποκεντρωμένης επεξεργασίας δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα ε, να προστατεύσουμε την Ευρώπη από πολλές απειλές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ας ανοίξουμε την συζήτηση. Ποιος, ποια μέλη θα ήθελαν το λόγο. Ο κ. Άλμπρεχτ, βλέπω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ στην κυρία Χολμάιερ. Μέχρι τώρα είχαμε μια πολύ καλή φιλική επικοδομητική συνεργασία και τη είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι' αυτό. Ένα-δύο ζητήματα ίσως θα ήθελα να ε, υπογραμμίσω εδώ και οδηγικά ότι δηλαδή καταρχάς ο προληπτικός ε, χαρακτήρας ε, θα πρέπει, ο χαρακτήρας της πρόληψης μάλλον θα πρέπει να προβληθεί ώστε να μην περιοριστούμε μόνο σε ένα κατασταλτικό μέτρο. Σε αυτό συμφωνούμε και με την εισηγητρία ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα σημαντικά μέτρα που θα θέλαμε μέσα στην οδηγία. Ζήτημα φυσικά είναι επίσης το πώς θα ή πού θα εντοπίσουμε τις προτεραιότητές μας. Εδώ συμφωνώ με τον κύριο Ενάντες Μπαταγιέ στην ε, έμφαση που θα εντοπισουμε τις προτεραιοτητες μας εδω συμφωνω με τον κυριο εναντες Μπαταγέ στην εμφαση που θα πρεπει να δοθεί και στους παραγωγούς αλλά και στους παρόχους των υπηρεσιών του ίντερνετ. Εκείνοι θα πρέπει να φέρουν τον κύριο ευθύνη για την εξασφαλίση της ασφάλειας στο ίντερνετ. Θα πρέπει δηλαδή στο στο δυνατό βαθμό να προστατεύουν ε, το δίκτυά τους έτσι ώστε να μην υπάρχει τρύπα ασφαλείας. Εξού και η παρατήρηση για την ε, ε, ανάγκη σε επενδύσεις και στην κατάρτιση και στον, ε, στη λειτουργία στο σχεδιασμό αυτών των συστημάτων είναι πολύ σημαντική για να έχουμε πρόληψη στο το δυνατόν. Επίσης, όπως είπε και η συγγετρία, είναι πολύ σημαντικό, το είπαμε και νωρίτερα, να μην περιοριστούμε μόνο στο να περιγράψουμε νέα ε, νέες εγκληματικές πράξεις, νέα δικήματα. Και ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουμε και το ζήτημα του κατά πόσον θα ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής ε, πράξεις προπαρασκευαστικές όπως ο εξοπλισμός σε hardware κτλ. Αυτά ίσως θα έπρεπε να τα δούμε με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα γιατί ίσως ε, διευρύνουμε υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής. και δεδομένου ότι θεωρούμε πως ε, η ε, πάροχοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα, θα πρέπει να φέρουν την κύρια ευθύνη και ότι θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση περισσότερο στην ε, πρόληψη και, στην δίωξη εκείνων όμως που πραγματικά ε, θέλουμε να πατάξουμε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην στρέψουμε τα πειρά μας εναντίον κάποιων οι οποίοι είναι ουσιαστικά αθώοι, δεν έχουν ευθύνη στην, ε, στις δυσλειτουργίες αυτού του συστήματος. Τα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν στο σύστημα αυτό. Αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσουμε ιδιαίτερω και εν των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Θέλει κανεί άλλο να λάβει το λόγο. Κύριε Μπρόνς, έχετε το λόγο. Μια ερώτηση μάλλον, όχι το σχόλιο. Η κυρία Χολμάιερ μας ενέφερε ως ε, ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί των ε, του ορισμού ε, λοιπόν η παράνομη δραστηριοτητων αναφερθηκε λοιπον ω παραδειγμα η εξασφάλιση πρόσβασης. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί στην οδηγία. Προφανώ θα μπορούσα να το έχω κοιτάξει και μόνο μου, δεν ήταν ανάγκη να διατυπώσω την ερώτηση. Αλλά ε, υπάρχει ενδεχόμενο φερρυπίν για επιβολή λογοκρισία ή για παρεμπόδιση κυκλοφορία των ηλεκτρονικών μηνυμάτων με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Ερνάντες. Άλλες ερωτήσεις. Δεν βλέπω να στεί κανείς άλλο το λόγο. Κύριε Ερνάντες, εσείς. Νομίζω ότι η, η ερώτηση αυτή απευθύνεται πιο πολύ προς την Κομισιόν που σύνταξε το κείμενο. Ε, εγώ, ερμηνεύοντας την πρόταση της Κομισιόν, θεωρώ πως η απάντηση είναι αρνητική. Αυτή όμως είναι η δική μου προσωπική άποψη. Άλλα σχόλια. ναι Then, no, comment. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από τα μέλη. Ίσως να αποτανθούμε προς το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλουν να πούν κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συνέταξε την πρόταση δεν γνωρίζει να υπάρχουν κάποιες άγνωστες λεπτομέρειες κυρίως όσον αφορά τη λογοκρισία ίσως σχετίζεται με μια συζήτηση που διεξάγεται όσον αφορά την άλλη οδηγία για την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Αλλά πρέπει να πω κάτι ξεκάθαρο για αυτή την περίπτωση. Ότι αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον μπλοκάρισμα έχει σχέση με τη λογοκρισία. Θέλουμε να μην μπορεί να υπάρξει είσοδο στις τοσελίδες εάν δεν μπορούν αυτές να αφαιρεθούν γρήγορα και να μπλοκάρονται οι εικόνες ε, παιδιών που είναι θύματα κατάχρηση ή είναι βιασμένα παιδιά. Δεν έχει σχέση με λογοκρισία όμω αυτό. Σα ευχαριστώ. Το Συμβούλιο. Η απάντηση είναι σαφώς όχι σε αυτή την ερώτηση. Δεν έγινε καμία απόπειρα στο Συμβούλιο να συμπεριληφθεί κανόνα περί λογοκρισία. Μιλάμε για την καταπολέμηση του εγκλήματο του κυβερνοχώρου και όχι για παράνομο περιεχόμενο του στο διαδίκτυο. Ελπίζω αυτό κάπως να σας καθησυχάζει. Ευχαριστώ. Η κυρία Χολμάιερ, η συγγήτρια. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχω διαβάσει πολλές φορές το κείμενο από πάνω μέχρι κάτω. Δεν υπάρχει πουθενά υπόνοια, η παραμικρή υπόνοια, συγκεκαλυμένη ημί για ε, λογοκρισία. Στόχος και μόνο αυτή της πρώτη οδηγία είναι η αντιμετώπιση των κακόβουλων επιθέσεων που έχουν σαν στόχο και ή και αποτέλεσμα την ε, πρόκληση ζημία σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και τον προσδιορισμό ελάχιστων προδιαγραφών με βάση τις οποίες θα αντιμετωπιστούν αυτού τύπου τα αδικήματα. Κάποιες έννοιες μάλιστα έχουν ε, διατυπωθεί κατά τρόπο ώστε μπορεί να μας φαίνονται κάπως ασαφείς ε, σε εμά και ίσως θα πρέπει ως εκ τούτου να συζητήσουμε τους ορισμούς πιο προσεκτικά ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι εννοούμε, ώστε να μην καταλήξουμε τελικά σε 27 διαφορετικές ερμηνείες αυτών των όρων, να μην έχουμε δηλαδή από κάθε κράτος μέλος ε, διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό πιστεύω δεν μπορεί να βοηθήσει ε, προσθέμενη αξία μπορούμε να έχουμε χάρη στο ευρωπαϊκό δίκαιο μόνο εάν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα με τον ίδιο όρο. Αυτό. Και επίσης θα μα απασχολήσει, πιστεύω, πάνω απ' όλα στο πλαίσιο αυτή τη οδηγία για το ποινικό δίκαιο, ε, σε ποιο βαθμό μπορεί να ε, συνδυαστεί η οδηγία αυτή περιπινικού δικαίου στο διαδίκτυο με μέτρα προληπτικά ή μήπως θα πρέπει να ε, προκύψει από ένα χωριστό κείμενο, από μια χωριστή έκθεση ε, στην Επιτροπή Μηχανίας Φερρυπίν. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε στόχο μας έχουμε ε, ένα πρόβλημα, ένα αδίκημα, να το ε, καταπολεμήσουμε, ένα φαινόμενο ε, εγκληματικό, να το καταπολεμήσουμε πρώτα προληπτικά και μόνο σε ίστατη λύση να θέσουμε σε λειτουργία της διατάξεις του ποινικού δικαίου, τη δίωξη, την εξέβρεση των ε, υπετίων και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η γενική μας νοοτροπία, αυτή είναι η θέση με βάση την οποία ορίζουμε ελάχιστε προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοινέ προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δούμε λοιπόν και από την Επιτροπή των, ε, της Βιομηχανίας και της, των Εξωτερικών ε, πώ θα ρυθμιστούν ή πώ θα αντιμετωπιστούν ορισμένα συστήματα όπω το cloud computing που αναφέραμε νωρίτερα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρέμβασή τη ανέφερε κάποια σημεία με τα οποία θα πρέπει να εμπλουτιστεί το κείμενο. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα κείμενο, μια οδηγία που θα πρέπει να ε, τύχει όσο το δυνατόν πιο δυναμική επεξεργασία, γιατί υπάρχουν τόσο ραγδαίε εξελίξει στον χώρο του ίντερνετ και τη τεχνολογία, πρέπει να είμαστε σε θέση να ε, εξασφαλίζουμε την προσαρμογή του δικαίου αυτού, ε, του νομοθετήματος αυτού, στις τελευταίες εξελίξεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Πρέπει να, έχουμε μια, ε, πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το κείμενο, δηλαδή αυτή η οδηγία, κατά τρόπο στο δυνατόν πιο ευέλικτο. Για το Συμβούλιο και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που είπε ο κύριο Άλμπρεχτ δηλαδή και θα μας απασχολήσει στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτά προς το παρόν στην πρωινή συνεδρίαση. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Να πάμε στο σημείο 17. Ευχαριστώ και Γιονάντες για την όλη παρουσίασή σας. Παρουσία στην Επιτροπή των Ελευθεριών, Μουσείων Ελευθεριών. Πολιτικών Ελευθεριών. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 17 όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και την παιδική πορνογραφία. Η κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη, συνάδελφο είναι εισηγήτρια. Το σχέδιο εκθέσεως τη εισηγήτριας, τη κυρία Αντζελίλη, υπευλήθη τον Ιανουάριο. Ακολουθήθηκε από ψηφοφορία προσανατολισμού το Φεβρουάριο. Και έτσι οι συγγήτρια και σκιώδει ε, εισηγητές ε, πήραν κάποιου προσανατολισμού για το ενδεχόμενο συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Διεξήχθησαν τον Μάρτιο τριμερείς διάλογοι και τον Απρίλιο και τον Μάιο και εξακολουθούν. Θα δούμε τώρα ποιες είναι οι εξελίξεις, θα μας τις αναφέρει η κυρία Αντζελίλη. Και μετά θα ακούσουμε τι έχει να μας πει το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Κυρία Αντζελίλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω απλώς μια ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες μας που αφορούν την οδηγία για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των ελίκων και την παιδική πορνογραφία. Το σημείο αναφοράς μας στις εργασίες μας ήταν η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του Λανζαρότε που αντιπροσωπεύει το σημείο αναφοράς, το πιο προχωρημένο σημείο αναφοράς στο νομοθετικό όσο αναφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων και την παιδική πορνογραφία θα ήθελα να τονίσω μόνο κάποια σημεία θετικά που συζητούμε, σημεία που επελύσαμε. εργαστήκαμε πολύ όσον αφορά τον ορισμό της παιδικής πορνογραφίας, επεξεργαστήκαμε τις ποινές, καταλήξαμε και σε κάποια συμφωνία που καθορίζει ποινές πιο κατάλληλες και που θα τιμωρεί και εκείνον που ε, εκμεταλλεύεται μια κυρίαρχη θέση, μια θέση εμπιστοσύνης, μια θέση επιρροής στους ανηλίκους που κα, ε, εκμεταλλεύεται το ευάλωτο χαρακτήρα του ανηλίκου όταν έχει φυσική ή ψυχική αναπηρία, το χάρη ο ανήλικος και ζητήσαμε πιο σημαντικές ποινές όσον αφορά ε, το, δίκημα, το έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας. Έχουμε εισαγάγει ένα στοιχείο που κατά την άποψή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει ήδη εισαχθεί στην οδηγία για το εμπόριο ανθρώπων δηλαδή κατάσχεση των αγαθών που σχετίζονται με το έγκλημα της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επεξεργαζόμαστε και τις απογορευτικές πίνες ούτω ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα εγκλήματα. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα, κυρίως μέσω ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τις καταδίκες για την εκμετάλλευση των ανηλίκων και την παιδική πορνογραφία, ούτω ώστε όποιος καταδικάζεται για αυτά τα εγκλήματα να μπορεί προσωρινά ή μόνιμα να μην μπορεί να ασκεί δραστηριότητες που οδηγούν σε μια τακτική επαφή αυτού του ατόμου με τους ανήλικους. Επεξαζόμαστε τις προδιαγραφές όσον αφορά το σεξουαλικό τουρισμό και όσον αφορά τις κυρώσεις που θα προβλέπονται και όσον αφορά τα μέτρα της πρόληψης. Προφανώς δεν είναι πολύ απλό αυτό, διότι αυτά τα δικήματα, τα εγκλήματα έχουν διεθνή χαρακτήρα Άρα θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα μέτρα που συνδέονται με την σχετική νομολογία. Δεν επεξεργαστήκαμε μόνο το θέμα της καταστολής αυτών των εγκλημάτων, αλλά και την πρόληψη αυτών και την προστασία των θυμάτων. Διότι αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της οδηγίας. Πολλά από αυτά τα εγκλήματα μπορούν ε, να αποφευθούν, να υπάρξει πρόληψη. Με, συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, των γονέων, των δασκάλων, των παιδιών, είναι πάρα πολύ σημαντική ανταλλαγή των πληροφοριών. Πρέπει να δημιουργηθεί και ένα σύστημα δικαιοσύνης υπέρ του παιδιού, να γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα του ανήλικου για να αποφύγουμε το δεδομένο φαινόμενο της να γίνεται διπλά θύμα το παιδί, δηλαδή να είναι αντικείμενο κατάχρηση, να είναι αντικείμενο εκμετάλλευση σεξουαλικής και μετά το παιδί ε, να γίνεται ξανά θύμα μέσω της δικαιοσύνης. Διότι ε, κρατούν πολλοί δίκες, παραδείγματο χάρη και σχετικές διαδικασίες, δεν υπάρχει επαρκή προστασία τη ιδιωτική ζωή του παιδιού και τα όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού, άρα το παιδί υποφέρει δύο φορές. Κλείνω αναφερόμενοι στο περίφημο άρθρο 21, το οποίο αναφέρθηκε και προηγουμένως, που αφορά όλα τα μέτρα, τα σχετικά με την εξάλληψη, με την διαγραφή του περιεχομένου του σχετικού με την παιδική πορνογραφία που είναι διαθέσιμο online. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ σειράς μέτρων, συνδυασμένων μέτρων που προβλέπουν πάνω απ' όλα την υποχρεωτική αφαίρεση κάθε παράνομου περιεχομένου που αφορά την παιδική πορνογραφία και διατίθεται online. Αλλά αυτή η αφαίρεση, η διαγραφή θα μπορεί να είναι δύσκολη, ίσως να απαιτεί μεγάλη χρονική περίοδο, διότι αυτές οι σελίδες μπορεί να εδρεύουν εκτός ένωσης. Χρειάζονται μέτρα που θα μπλοκάρουν την πρόσβαση. Έχουμε εμπειρία στην Ευρώπη σημαντική όσον αφορά αυτό το θέμα. Είμαστε τα κράτη-μέλη μας σε θέση, υιοθετώντα διάφορα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, είμαστε σε θέση και να παρεμβαίνουμε όσον αφορά την αφαίρεση, την έγκαιρη αρκετά ταχεία του παράνομου περιεχομένου, αλλά και έχουμε και συστήματα που μπορούν να αποκλείσουν την πρόσβαση, που είναι αποτελεσματικά συστήματα μπλοκαρίσματος με τη συνεργασία και με τα διάφορα δίκτυα των παρόχων των υπηρεσιών ίντερνετ. Όσον αφορά το μπλοκάρισμα και την αφαίρεση, δεν μιλάμε ποτέ για λογοκρισία όταν μιλάμε για αυτά τα μέτρα. Ε, μιλάμε για την παιδική πορνογραφία. Προφανώς εμείς έχουμε ορίσει τι αποτελεί, τι είναι αυτή η παιδική πορνογραφία. Στο άρθρο 2 υπάρχει ορισμός, σαφέστατος, αδιαμφισβήτητος δεν μιλάμε για διαφημίσεις, ξέρω εγώ, που θα μπορούσαν ε, να είναι κάπως προκλητικές, πονηρές, θα μπορούσαν ε, να έχουν κάποιες αναπομπές εξοκαλικά ε, θέματα. Δεν μιλάμε αυτού του είδους την ενημέρωση, την επικοινωνία. Δεν ανεφερόμαστε στην ελευθερία της σκέψης. Μιλάμε μόνο για εικόνες τις οποίες διαπράζεται ένα αδίκημα σαφές, προφανές αδίκημα που αφορά είναι σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού, είναι δύο αδίκημα, είναι αδίκημα που, όλοι, που τιμωρούνται από όλου ποινικού κώδικες, όχι μόνο ευρωπαϊκούς, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Όταν μιλάμε για φέρεση της ή μπλοκάρισμα, μιλάμε για φέρεση του περιεχομένου ή μπλοκάρισμα του περιεχομένου, μπορεί να είναι εικόνες, ταινίες, βίντεο κλιπ, Αφαίρεση λοιπόν και μπλοκάρισμα από εικόνες όπου σαφέστατα και αδιαμφισβήτητα έχουμε ε, βία πράξη κατά του παιδιού, έχουμε ε, ε, σεξουαλική εκμετάλλευση του ανηλίκου. Είναι μια εικόνα που δεν μπορεί να ερμηνευτεί, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας προσέγγισης διαφορετικής όσον αφορά τα πολιτισμικά. Είναι ένα δίκημα που καθορίζεται σαφώς ένα έγκλημα που αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας σαφώς. Η ελευθερία της έκφρασης ή ενδεχόμενη λογοκρισία όσον αφορά ε, το θέμα αυτό που σχετίζεται με την αφαίρεση του περιεχομένου, το μπλοκάρισμα του περιεχομένου δεν μπορεί να υφίσταται διότι μιλάμε για πάρα πολύ σαφή εγκλήματα. Πιστεύω ότι τα είπα όλα, όπως υπενθύμισε και ο Πρόεδρος, ε, εργαζόμαστε προσπαθώντας να ψηφίσουμε ε, το κείμενο τον Ιούνιο ούτως ώστε μετά να το υποβάλουμε στην Ολομέλεια, στη Σύνοδο τέλους Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Όμως δεν προτιθέμεθα να κάνουμε συμβιβασμούς προς τα κάτω. Εάν χρειάζεται περισσότερο χρονικό διάστημα και ενεργαστούμε περισσότερο θα το κάνουμε αυτό και μετά ε, θα αναβάλουμε αργότερα την ψηφοφορία. Ευχαριστώ κυρία Αντζελίλη και τώρα ας ακούσουμε τι έχει να πει πρώτα το Συμβούλιο πριν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Προεδρία ίσως ε, θέλει να παρέμβει. Ορίστε. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια και παίρνω το λόγο για δεύτερη φορά, θα παραλείψω τις εισαγωγές. Θα ήθελα να πω στην ουσία ότι με πολύ μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε σημαντική πρόοδο και ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις αυτές και ελπίζουμε να καταλήξουμε κατά τη διάρκεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας ακόμη σε συμφωνία μαζί σας. Αυτό που σημειώνουμε είναι η αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην υπόθεση αυτή. Πρόκειται για μια από τις ε, μεγάλες προκλήσεις για το παρόν και το μέλλον. Η δε Ουγγρική Προεδρία είναι στρατευμένη στον αγώνα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και έχει αναλάβει εντατικές συζητήσεις με την εισηγήτρια και τους συναδέλφους της. Ελπίζουμε ότι θα εξασφαλίσουμε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό. Ασφαλώς αντιλαμβανόμαθα ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση. Έτσι συμβαίνει πάντα στις πραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έτσι για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και να εκφράσω την ευχή ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία στο εγγύς μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Γιάκο την Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Πολύ σύντομα, διότι θα ήθελα και εγώ να εκφράσω εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκτίμηση των προσπαθειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των στόχων του. Όντω, έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα ολιστικό ε, μέσο, εργαλείο και στην ουσία προσφέρουμε προσθέμενη αξία ως προς συγκεκριμένους ορισμούς πολλών και διαφορετικών αδικημάτων με την δυνατότητα προσφέρει ένα τέτοιο ολιστικό έγγραφο να μπορούμε να αποτρέψουμε υποτροπιασμό, ο οποίος διαπιστώθηκε στην αποτρόπια εκείνη υπόθεση Φουρνιρέ Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί αυτή η οδηγία να δώσει σημαντική προσθέμενη αξία σε κάθε μέτωπο της μάχης κατά της παιδικής πορνογραφίας. Ωραία. Σύντομα ε, και λιτά θα μπορούσαμε να ε, ξεκινήσουμε τη συζήτηση, αλλά η ηλεκτρονική πλειοψηφία είχε προγραμματιστεί για τις 10, οπότε δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να περάσουμε στην ψηφοφορία πολύ γρήγορα, γιατί κάποια μέλη πρέπει να φύγουν, έχουν άλλες ε, υποχρεώσεις. Παρακαλώ πολύ να έχετε έτοιμες τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Αν δεν τις έχετε, στείλτε κάποιον να τη φέρει. Ε, θέλετε... Ο κ. Σκύρκοπ ε, της διαδικασίας. Κυρία Βίξτρομ, έχετε το λόγο. Συζητάμε την έκθεση Αντζελίλη περνάμε στην ψηφοφορία. Όχι, συζητάμε την, ε, την έκθεση Αγγελίλη. Ε, απλά είπα ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει για τις ε, ε ψηφοφορίες και αυτό είναι πρόβλημα για ορισμένα κράτη-μέλη γιατί ε, ορισμένα από αυτά έχουν άλλες υποχρεώσεις και πρέπει να τελειώνουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της. Θα μπορούσαν παρακαλώ τα μέλη να καθίσουν και να είναι ήσυχα γιατί έτσι δυσκολευόμαστε πολύ. Ναι, ναι, παρακαλώ πολύ ησυχία, λέει ο Πρόεδρος, παρακαλώ πολύ ησυχία. Ε, ελπίζω κύριε Αντζελίλη να ακούσατε ότι σας ευχαρίστησα για την προσήλωσή σας σε αυτό το ζήτημα. Φτάσαμε σε καλούς συμβασμούς σε ορισμένα δύσκολα πολιτικά ζητήματα. Και τώρα συζητάμε, συνεχίζουμε τη συζήτηση σε πιο τεχνικά ζητήματα για να ξεκαθαρίσουμε όλη την έκθεση για να πάει κάθε τροπολογία εκεί ε, στο, στη θέση της. Η πολιτική εστίαση είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο ίντερνετ. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση όμως. Θα πρέπει να επωφεληθούμε της ευκαιρίας για να καταπολεμήσουμε την ε, κακοποίηση εκεί που υφίσταται, στην καθημερινή ζωή. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που βλέπουμε στο ίντερνετ είναι ένας ε, καθρεφτισμός αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Το ίντερνετ δεν είναι ένας ξεχωριστός χώρος όπου όλα επιτρέπονται. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα εγκλήματα και στο ίντερνετ. Αλλά αυτό που είναι παράνομο στην πραγματική ζωή θα πρέπει να θεωρείται παράνομο και στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε να νομοθετούμε για το ίντερνετ με τρόπο που δεν έχουμε στην πραγματική ζωή. Θα χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση και ελπίζω πραγματικά ότι θα επιτύχουμε αποτελέσματα με αυτήν την έκθεση. Ελπίζω ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά για να το κλείσουμε κατά τη διάρκεια της Ουγγλικής Προεδρίας το ζήτημα αυτό, χρειάζεται να πείσουμε το Συμβούλιο για το άρθρο 21. Θα πρέπει να γίνει δεκτή το συμβαστικό κείμενο του Κοινοβουλίου που καθιστά σαφές πως ε, τα κράτη-μέλη θα αποσβήνουν, θα διαγράφουν ότι και μπορούν θα διαγράφουν ενώ μπορούν να μπλοκάρουν. Shall delete may block. Νομίζω ότι για να καταλήξουμε σε συμφωνία πρέπει να γίνει δεκτός αυτός ο συμβασμός. Ευχαριστώ. Now, Mr. Kirchhoff. Κύριος Εν συντομία, γιατί ξέρω ότι πρέπει να ψηφίσουμε, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Αντζελίλη και συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Wickstrom για το ίντερνετ. Ε, ο συντάκτης της αρχικής μας έκθεσης εδώ και πολλά χρόνια για την εκμετάλλευση παιδιών μέσω του ίντερνετ δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να ξεχνάμε τα όσα έχουμε πει. Δύο σχόλια. Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες. Καταλαβαίνουμε ότι οι νομοθέτες σε όλη την Ευρώπη χρειάζεται να έχουν κάποια ταξινόμηση, αλλά να θεωρούμε παιδί οποιονδήποτε είναι κάτω από 18 δημιουργεί δυσκολίες στην ταξινόμηση. Ε, κάθε χώρα έχει τη, τη δική της πολιτική κατανόηση των πραγμάτων. Άλλη είναι η βλάβη που παθαίνει ένα παιδί 14 ετών, άλλη η βλάβη ενός παιδιού 6 ετών. Επίσης υπάρχει μια, ένα κεφάλαιο για την πρόληψη, ε, αλλά θα ήθελα να γίνει πιο λεπτομερές. Καλές οι κυρώσεις, καλές οι ποινές, αλλά το κλειδί είναι η πρόληψη. Και θα έπρεπε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Τέλος, για το άρθρο 19, τα δικαιώματα των θυμάτων. Ε, θα μπορούσαν όλα αυτά να συμπεριληφθούν και στο πακέτο των δικαιωμάτων των θυμάτων, ε, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην αλληλεπικαλυφθούμε γιατί μπορεί να δημιουργηθούν παρανοήσεις. Ευχαριστώ. Ξέρετε κατά τα άλλα η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Αντζελή, το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Ευχαριστώ και ο Σάλμπρεχτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα στην εισηγήτρια για τη δουλειά τη την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι, το κατέστησε φεσκή κυρία Ρίξ ότι στόχος μας κοινό είναι η καταπολέμηση της ε, εκμετάλλευσης των παιδιών. Και μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το χώρο της ε, συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών ή δικαστικών αρχών, και ταυτόχρονα θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει εμεί ω βουλευτέ το θέμα αυτό να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, όχι δηλαδή μόνο συγκινησιακά, αλλά με ψυχραιμία και να ασκήσουμε πιέσεις εκεί όπου ακριβώς θα είναι χρήσιμο για να έχουμε πιο καλό αποτέλεσμα. Έχουμε κάνει πολλές συμβαστικές τροπολογίες, έχουμε καταλήξει σε πολλούς συμβασμούς εδώ στην Επιτροπή μας και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι έχουμε μια σαφέστατη θέση στην Επιτροπή μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία. Καταρχάς το ζήτημα των ορισμών, διότι θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να μιλάμε όπως κάναμε μέχρι τώρα για παιδική πορνογραφία, αλλά για υλικό που δείχνει εκμετάλλευση παιδιού μας του ίντερνετ. Πορνογραφία σημαίνει ε, ή μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μια αποδεκτή ή για μια συνενετική πράξη, πράγμα το οποίο αποκλείω βέβαια ε, απολύτως δεν υπάρχει καμία σχέση με την συνένεση στην περίπτωση της παιδικής πορνογραφίας. Πρόκειται για κατάχρηση παιδιών, για εκμετάλλευση σεξουαλική παιδιών, για εγκληματική ενέργεια. Αυτό πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφέ. Επίση, πολύ σημαντικό για μένα είναι το να δούμε όλη αυτή η συζήτηση ω προ ε, το υλικό που προκύπτει από σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο ίντερνετ. Ε, έχουμε καταλήξει μια συμβαστική πρόταση πολύ καλή, την οποία υποστηρίζουν τέσσερις πολιτικές ομάδες εδώ στην Επιτροπή μας και η οποία λέει ότι η διαγραφή του περιεχομένου αυτού πρέπει να αποτελεί την κατά προτεραιότητα ενέργεια που θα αναλευθεί σε περίπτωση ε, παρουσίας τέτοιου ε, υλικού στο ίντερνετ. Πρέπει να φροντίζουμε δηλαδή το υλικό αμέσως να διαγράφεται, να κατάσχεται ούτως υπήν εντός εισαγωγικών, να απομακρύνεται από τον δικτυακό χώρο στον οποίο εντοπίζεται. Έτσι ώστε η ιδέα της συνεργασίας να μην ε, καθιστά την αντιμετώπιση του αδικήματος αυτού πιο ασαφή ή να μην την ε, νερώνει εντό εισαγωγικών. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία με βάση αυτή την ε, νέα νομοθεσία να μπορέσουμε να έχουμε κοινού κανόνες και προδιαγραφές για την ε, αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων, για την αστυνομική συνεργασία, για τη δικαστική συνεργασία, ώστε να μην υπάρχει η εντύπωση ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιωτικό ή ιδιωτικού δικαίου που ρυθμίζεται ιδιωτικά. Πρόκειται για ένα ποινικό ζήτημα, το αντιμετωπίζουν οι κρατικές αρχές και γι' αυτό θέλουμε το Συμβούλιο να προχωρήσει όχι στον αποκλεισμό της πρόσβασης αλλά στην διαγραφή, να συμφωνήσει δηλαδή στη διαγραφή του υλικού αυτού. Ευχαριστώ η κυρία Μποσκούρτ παρακαλώ, σύντομα όμως γιατί ξέρετε ότι μας περιμένουν οι συνάδελφοι για την ψηφοφορία. Ναι, το ξέρω πρέπει να ψηφίσουμε. Έχω όμως και εγώ κάτι να πω και είναι πολύ σαφή αυτό που έχω να πω. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, ε, δεν νομίζω ότι αξίζει να το συζητάμε τόσο σύντομα και τρία λεπτά μόλις πριν τις προφορίες. Πολύ σύντομα λοιπόν. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει όλη αυτή την υπόθεση στην ε, παρουσίασή της μας μίλησε για τη σημασία της πρόληψης, συμφωνώ απολύτως, αλλά έχω να διατυπώσω και μια συγκεκριμένη ερώτηση σε σαφείς όρους στην πρόληψη και προκειμένου να αποφύγουμε ένας εγκληματίας ο οποίος έχει ε, καταχραστεί παιδιά ε, κατά τρόπο σεξουαλικό ή άλλον. Να αποτρέψουμε λοιπόν αυτός ε, ο εγκληματίας ε, να διαφύγει και να περάσει σε άλλο κράτος μέλος όπου θα ξαναρχίσει τις εγκληματικές δραστηριότητες, θα ήθελα, και το έχω ζητήσει μια τροπολογία, ένα μητρό πανευρωπαϊκό, το οποίο θα επιτρέπει να εντοπίζεται ο παιδεραστής ή ε, ο υπέτειος τέτοιων αδικημάτων εις βάρος των παιδιών, ώστε να τους ε, χαρακτηρίζουμε τροποντινά και να μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη των ίδιων πράξεων. Ε, έχει γίνει δεκτή από την Επιτροπή αυτή η τροπολογία. Επίση, γνωρίζω ότι και κάποιε από τι χώρε μέλη στο Συμβούλιο, όπω η δική μου, επί παραδείγματι, έχουν δεχθεί την ιδέα αυτή. Θα ήθελα να ρωτήσω ω προ τη διαδικασία, εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί με ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό και θα ήθελα να περάσει. Ευχαριστώ, κύριο Μπρόν. Ε, ήμουν παρόν στην ακρόαση την, ε, το, που έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Τα πρώτα λεπτά τουλάχιστον ήμουν και ο μόνο, νομίζω και ε, ήταν παρόντες και εκπρόσωποι των θυμάτων. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώμη τους. Ε, πρώτον, διαφωνούν με τη χρήση του όρου παιδική πορνογραφία, όπως είπε ο κύριος Άλμπρεχτ. Δεύτερον, διαφωνούσαν με το μπλοκάρισμα των ιστοσελίδων αντί για την αφαίρεσή τους, ως υποκατάστατο της αφαίρεσής τους. Ασφαλώς και το μπλοκάρισμα δεν είναι υποκατάστατο, ε, αλλά από ό,τι φαίνεται προτείνουν ε, μάλλον φαίνεται να πιστεύουν ότι ε, δεν είναι καλύτερο το μπλοκάρισμα το να μην κάνουμε και τίποτα. Ε, Επίση, μετά την ακρόαση, ε, μίλησα με, με έναν εκπρόσωπο του κλάδου της ε, τεχνολογίας των πληροφοριών και μου είπε ότι είναι δυνατόν τεχνικά ε, άνθρωποι που παρέχουν τέτοιου είδους υλικό να αποτελούν κομμάτι ενός νόμιμου site. Αυτό συνέβη κιόλας με κάποιους ε, ε, πολύ τίμιους και ε, επαγγελματίες ε, των οποίων ένα κομμάτι του site κατά κάποιο τρόπο τεχνικά που εγώ αγνώ τεχνικά πώς έγινε ε, καταλήφθηκε από ένα site παιδικής πορνογραφίας. Κυρία Ιντβέλτ, θα μπορώ, μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Η συζήτηση έχει γίνει, έχουμε υιοθετήσει μια θέση, είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξαναγίνει όλη η συζήτηση. επιθυμούμε ε, η ε, η συγγήτριά μας να προωθήσει τις απόψεις μας ε, στον τριμερή διάλογο. Στη θέση μας υπογραμμίζουμε την ανάγκη διαγραφής απόσυρσης του περιεχομένου και όχι του μπλοκαρίσματος. Αυτό θα ήθελα η, η συγγήτρια να προωθήσει σε απόψή μας. Κυρία Αντζελίλη, Τελειώνουμε, κλείνω πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας για τις ερωτήσεις, για τα σχόλια που ακούστηκαν. Δεν έχω πολύ χρόνο, συνεπώς θα είμαι πολύ σύντομη στην απάντησή μου. Είμαι πεπισμένη ότι σε ό,τι φορά το άρθρο 21, ε, το κοινοβούλιο ήταν πολύ σαφής, σαφές. Ε, στόχος μας είναι η απόσυρση, η διαγραφή του περιεχομένου. Το μπλοκάρισμα θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν είναι δυνατόν ή καθώς ο χρόνων δεν είναι δυνατή η διαγραφή του περιεχομένου. Γιατί η διαγραφή μπορεί να καθυστερήσει μέρες, εβδομάδες ή μήνες. Συνεπώς είναι λογική αυτή η άποψή σας. Παρακαλώ λοιπόν να διαβάσετε τα επίσημα έγγραφα. Προσθέσαμε μερικά πράγματα γιατί ακούσαμε την Ευρωπόλ, την Ιντερπόλ κλπ. Ενημερωθήκαμε, συλλέξαμε όλες τις εμπειρίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι εμπειρογνώμονες μας είπαν, ο στόχος είναι η διαγραφή του, περιεχο... του παράνομου περιεχομένου. Όπως ακριβώς γίνεται και στην πραγματικότητα. Αλλά εν αναμονή της διαγραφής, αν αυτή η διαγραφή δεν μπορεί να γίνει αμέσως, πρέπει να μπλοκάρουμε το περιεχόμενο. Ο τελικός στόχος όμως είναι η διαγραφή. Αν χρειαστεί ε, ένα χρονικό διάστημα, δύο, τρεις μέρες, μία εβδομάδα για να γίνει η διαγραφή, για να αποσυρθεί από το ίντερνετ αυτό το περιεχόμενο που αποτελεί προϊόν εγκλήματος, ε, αν καθυστερήσει, καθ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περίοδου μπορούμε να μπλοκάρουμε το περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει ήδη στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες. Σε ό,τι αφορά τους ορισμούς, παιδική πορνογραφία, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα, όλες τις διεθνείς συμβάσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεταγράψουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και συμβάσεις όπως η Σύμβαση του Λανσαρότε, ε, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη και δεν πρέπει να επιτρέψουμε το νομικό το νομοθετικό πλαίσιο να χάσει την ομοιογένειά του και τη συνέπειά του. Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο κατάλογο και το σύστημα έκρηση, ε, συμφωνώ, αλλά το πιο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη υποχρεωτικά να μοιράζονται τις πληροφορίες που διαθέτουν. Αυτό δεν ισχύει, αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνει η χώρα. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι θα πρέπει να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες έτσι ώστε τα μέτρα να έχουν αποτέλεσμα. Το Κοινοβούλιο θα δώσει μάχη για να το πετύχει αυτό. Γιατί είναι σημαντικό το σύστημα να είναι λειτουργικό έτσι ώστε όποιος διαπράττει τέτοιου είδους αδικήματα να είναι γνωστός από όλου. Σταματάω εδώ γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρόεδρε. Ε, ένα μόνο πράγμα θα πω. Κανένας από εμά δεν έχει ε, προκαταλήψεις. Εγώ χρησιμοποιώ το ίντερνετ, η κόρη μου από τεσσάρων ετών χρησιμοποιεί το ίντερνετ, γιατί είναι κάτι το μοναδικό. Εγώ όταν ήμουν μικρή, 5-6 χρονών δεν είχα δυνατότητα να έχω πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν υπήρχε τότε. Ε, είμαι υπέρ τη ελευθερία έκφραση, είμαι υπέρ τη δημοκρατία, Όλα αυτά είναι πολύ θεμελιώδη. Αλλά αν, όταν λαμβάνει η χώρα ένα αδίκημα θα πρέπει να παρεμβαίνουμε. Πρόεδρο, ευχαριστώ κύριε Αντζελίλη. Νομίζω ότι συζητήσαμε επαρκώ το θέμα. ο τριμερής διάλογος θα συνεχιστεί έτσι ώστε να καταφέρουμε να ψηφιστεί το θέμα τον Ιούνιο ε, στην Επιτροπή μας και αργότερα στην Ολομέλεια. Ε, κύριε Άλμπρεχτ, για τη διαδικασία. Θα ήθελα μόνο να καταστώ σαφές ότι τη θέση του Κοινοβουλίου και τη στάση του στις λοιπές διαπραγματεύσεις θα την καθορίσει το κείμενο πάνω στο οποίο έχουμε συμφωνήσει και όχι η διατύπωση την οποία επέλεξε να χρησιμοποιήσει τώρα η εισηγήτρια. Η παρεμπόδιση πρόσβασης δεν είναι το ελάχιστο αποδεκτό για το πρόβλημα αυτό για μας. Δεν έχει γίνει αποδεκτό αυτό. Ω εναλλακτική σε σχέση με την διαγραφή. Μόνο όταν αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατή η διαγραφή και υπό ορισμένε συνθήκε που έχουμε ε, διατυπώσει, μόνο τότε μπορεί εναλλακτικά να γίνει δεκτή ω λύση η παρεμπόδιση πρόσβαση. Αυτό ήθελα να καταστεί απόλυτα σαφές. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άλμπρεχτ, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο είπατε, αλλά θα σα υπενθυμίσω ότι ε, όταν σηκώνουμε τα χέρια μας και τα σταυρώνουμε για να ζητήσουμε παρατήρηση επί του κανονισμού, ε, πρέπει να τηρούμε και τον κανονισμό τον ίδιο, γιατί διαφορετικά το να κάνουμε πολιτικές τοποθετήσεις ε, παραβιάζεται, τον ίδιο, παραβιάζεται ο ίδιος ο κανονισμός. Παρακαλώ λοιπόν. Αλλιώς θα σηκώνει το καθένας να παίρνει το λόγο και δεν θα μπορούμε να σταματήσουμε ποτέ αυτό το φαύλο κύκλο. Τώρα θα, με, θα υποχρεωθώ να δώσω το λόγο και πάλι στην εισηγητρία για τη διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων, ώστε να επανέλθουμε για τη ψηφοφορία. Κύριε Αντζελίλη, μια κουβέντα μόνο. Προφανώ εγώ εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο και ε, προασπίζω με τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Συνδυάζω δε όλες τις συμβαστικές, ακολουθώ δηλαδή όλες τις συμβαστικές τροπολογίε. Εδώ δεν έχω να κάνω, δεν εκφράζω ε, προσωπική μου θέση. Στου και ηγητές ναι μπορώ να την εκφράσω, αλλά όχι στον τριμερή διάλογο ενώπιον του Συμβουλίου και τη Επιτροπή, Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ιδάλλως ε, δεν μπορώ ε, να ισχυριστώ ότι επιτελώ το έργο μου όπως ε, οφείλω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να επενθυμίσω σε όλους τους βουλευτές ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουν το κείμενο και όταν γίνονται παρεμβάσεις επί της αρχής και δηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα από κάποιους, ενδεχομένως αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν διαβάσει προσεκτικά όλο το κείμενο και τις αιτιολογικές σκέψεις συμπεριλαμβανόμενες. Επίσης λοιπόν θα ήθελα να πω ότι για τον κύριο Άλμπρεχτ ότι προφανώς δεν έχει διαβάσει με την προσοχή που όφιλε το κείμενο. Ο πρόεδρος προφανώς θα το διαθέσουμε το κείμενο, ε, θα το, δημοσιε... θα το κυκλοφορήσουμε αλλά η παρατήρηση ασφαλώς είναι θεμητή ε, στο βαθμό που μπορεί κανείς να την εκφράσει εν ευθέτω χρόνο μέσα από την ψηφοφορία. Από εκεί πέρα θα δούμε πώς η ε, ε, διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο θα εξελιχθούν και βέβαια ποιε τη θα κρατηρήσει ο καθένα στην ψηφοφορία. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία γιατί έχουμε αυτό το θέμα πρώτα και μετά έχουμε και την Επίτροπο Ρέντινγκ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Παρακαλώ ήσυχη. Ας ξεκινήσουμε. Αλλά επιτρέψτε μου πρώτα δύο ανακοινώσει. Πρώτον, Η έκθεση για τον συνολικό κώδικα Σέγγεν ε, ε, κατοχυρώθηκε στον κύριο Παπα-Νικολάου. Δεύτερον, προθεσμία για τις τροπολογίες για την έκθεση του κύριου Κοέγιο για το μηχανισμό αξιολόγησης Σέγγεν ε, ήταν, είναι σήμερα στις 12. Ο εισηγητής έλαβε αιτήματα να παραταθεί αυτή η προθεσμία. Συμφωνεί με αυτά τα αιτήματα, οπότε η καινούργια προθεσμία είναι μέχρι την 5η, 26 Μαΐου, 5 το απόγευμα. Μέχρι την 5η, 5 το απόγευμα μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες. Ψηφίζουμε. Δύο γνωμοδοτήσεις. Έχετε ελπίζω τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Πρώτη γνωμοδότηση είναι αυτή της κυρίας Μπλίνκεβισιούτε. Περί, την κινητικο... περί της κοινωνικότητας των ε, εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογίες 6 και 7 καταπίπτουν, 8 καταπίπτουν, 9 καταπίπτουν. Δεύτερη συμβαστική λύση, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε 15, χωριστή τροπολογία, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, συγγνώμη. Το ελέγχουμε. Δεύτερο τμήμα. Ελέγχουμε. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 24 υπέρ, 24 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε και πάλι ηλεκτρονικός, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη 16. Κλείνει η ψηφοφορία. 24 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στη 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Και πάλι χωριστή ψηφοφορία. Μόνο το πρώτο τμήμα. Καταρχήν το πρώτο τμήμα της 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 5. Συμβαστική πρόταση 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε. Κάποιες καταπίπτουνε. Περνάμε κατευθείαν στην 33. Προφορική τροπολογία του κ. Κίρκοπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας το, ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. «23 υπέρ 21 κατά». Εγκρίνεται. Καλά κάναμε και ελέγξαμε όμως. «34 υπέρ» κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές ας, ας ελέγξουμε για την 35 άρχεται η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία «25 υπέρ 18 κατά» και πάλι εγκρίνεται. Ναι. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Τι ήταν, υπέρ ή κατά. 26 υπέρ, 19 κατά. Λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 δεν καταπίπτει. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 με προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 ο, και 46 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πολύ, κατά πολύ. Τροπολογία, ε, συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 δεν έχει καταπέσει, δεν καλύπτεται από το συμβαστική 7, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 53, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα, αιτιολογικέ παραγράφη της έκθεση. έκθεση. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου. Όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Now, we proceed to the second opinion on the vote, which is the opinion... Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, γνωμοδότηση για την εντολή για τον τριμερή διάλογο για το σχέδιο προπολογισμού του 2012 η συγγήτρια συνάδελφος η κυρία Κέλλερ, η Φραντσίσκα Κέλλερ. Πάμε αμέσως στις τροπολογίες. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται απορρίπτεται ας γίνει έλεγχος για το δεύτερο τμήμα έλεγχος ξεκινάει η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 7 τι έχουμε 27 κατά 17 υπέρ απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές ας γίνει έλεγχος για τη 13 ξεκινάει ο έλεγχος ηλεκτρονικό. ηλεκτρονικός Τέλος. 24-21 εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ας κάνουμε έναν έλεγχο για την 11 έλεγχος για την 11 ξεκινάει τέλος απορρίπτεται απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τι είπατε να ελέγξουμε τη 12 νομίζω ότι απορρίπτεται ας γίνει έλεγχος για τη 12 έλεγχος για τη 12 έλεγχος 12 ξεκινάμε τέλος απορρίπτεται τροπολογία η προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές το ίδιο εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές ας γίνει έλεγχος αυτή τη φορά έλεγχος για την 18 18 έλεγχος που ξεκινάει τώρα τέλος 21 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται 19 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές αναφορές, αιτιολογικές σκέψεις. Ένα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο ως ετροποποίηθη. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 42 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαίρουμε λοιπόν την κυρία Κέλλερ. We have now... Τώρα έχουμε σημείο 20 τον διαθρωμένο διάλογο με, το, με τον Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια, την κυρία Ρέιντινγκ, σχετικά με την εκτέλεση του Προγράμματος Εργασία Επιτροπής για το 2011 και την προετοιμασία του μελλοντικού πρόγραμμα της εργασίας επιτροπής για το 2012. Ε, είναι ανταλλαγή απόψεων σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει πριν τον Ιούνιο κάθε επίτροπος να υποβάλει το ποια είναι η κατάσταση, να ενημερώνει την κατάσταση του νεστότος προγράμματος του 2011 και τι προβλέπεται όσο αφορά το πρόγραμμα εργασίας για το 2012. Καλωσορίζουμε την Αντιπρόεδρο, την κυρία Επίτροπο, την κυρία Ρέντινγκ. Καλώς ήρθατε σήμερα. Καλή σας μέρα. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το σημείο 20 για το διαθρωμένο διάλογο, ακούγοντας την κυρία Ρέντινγκ και μετά θα ξεκινήσει η ανταλλαγή των ε, απόψεων. Σας παρακαλώ όμως, αν έχετε την καλοσύνη, εσείς στην αίθουσα να κάνετε λίγη ησυχία και να δώσουμε το λόγο στην Επίτροπο την κυρία Ρέντιν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπω στο βασικό μας θέμα, διότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ε, θα ξεκινήσω με την ετήσια έκθεση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αρχές Απριλίου παρουσίασα την πρώτη ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της χάρτας. Ένας από τους στόχους της εκθέσεως ήταν η διευκόλυνση των συζητήσεων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της χάρτας και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που αυτή την εβδομάδα το Συμβούλιο υιοθέτησε τα συμπεράσματα του και το σημαντικότερο ότι υπογράμμισε τις ευθύνες που έχει για την εφαρμογή της χάρτας και για την ενημέρωση των πολιτών περί του πεδίου εφαρμογής της χάρτας. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα έκανε τώρα το Συμβούλιο και θέλω να ακούσω και εσείς τι έχετε να πείτε, τι έχει να πει το Κοινοβούλιο, η συγγήτρια, η κυρία Φλασίκο Μπένοβα, ούτω ώστε και το Κοινοβούλιο να συμβάλλει στη συζήτηση. Κοινό μας καθήκον είναι να ενημερώσουμε το ευρύτερο κοινό για την κατάσταση που δημιουργείται με τη χάρτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ, έχουμε συνεδρίαση, ακούμε την Αντιπρόεδρο, την κυρία Ρέντινγκ. Σας παρακαλώ λοιπόν οι παριστάμενοι να κάνουν ησυχία για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει η κυρία Ρέντινγκ. Το Συμβούλιο έκανε τη δουλειά του. Περιμένω τώρα να δω ποιες θα είναι οι εργασίες του Κοινοβουλίου επί του θέματος και όλοι μαζί έχουμε το καθήκον να ενημερώσουμε το ευρύτερο κοινό όσον αφορά που, για που ισχύει η χάρτα και που όχι. 4.000 επιστολές έλαβα, ξέρετε, πέρσι όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα τρία τέταρτα αυτών αφορούσαν υποθέσεις εκτός της, του πεδίου εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό ε, το θέμα αυτό και θα οργανώσουμε ένα σεμινάριο με συμμετοχή των ε, διαφόρων εθνικών φορέων των, ε, που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών, συμμετοχή του, Εθνικού, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δούμε πώς μπορούμε να, δώσουμε, να ενημερώσουμε τους άλλους αρμόδιους εθνικούς φορείς για τις διαμαρτυρίες που αφορούν θέματα που δεν άπτονται της χάρτας, διότι οι πολίτες δεν ξέρουν σε ποιον απευθυνθούν και έχουν πρόβλημα πολύ συχνά. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο τόσο ώστε ε, αυτομάτως να παίρνουν ε, οι πολίτες απαντήσεις από τους αρμοδίους φορείς. Λοιπόν, το φθινόπωρο θα διοργανωθεί ένα σεμινάριο σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ένταξη των Ρωμά ε, βάσει της εκθέσεώς σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την στρατηγική, για τις στρατηγικές εθνικές για την ένταξη των Ρωμά. Ε, συζητήθηκε αυτό στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης από τους Υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων, από τους Υπουργούς Παιδείας. Συζητήθηκε επίσης και τη Δευτέρα θα στο Συμβούλιο ΓΑΚ των Γενικών Υποθέσεων και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρωμά εγκρίθηκε, αυτό είναι το θετικό. Ε, συμπεράσματα έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο και θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου ούτως ώστε βάσει αυτών οι εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρώμα θα ε, καταρτιστούν και θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2011 και μαζί με τον συνάδελφό μου τον κύριο Άντορ θα έρθω ξανά εδώ το 2012 να σας ενημερώσω ε, περί των εθνικών στρατηγικών. Διαδικαστικά δικαιώματα ολοκληρώσαμε το θέμα του δικαιώματος διερμηνίας και μετάφρασης σε ποινικέ υποθέσεις, χάρη στη βοήθεια της κυρίας Σίπελ, της εισηγήτριάς σας, η οδηγία για το δικαίωμα της ενημέρωσης σε ποινικέ υποθέσεις έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο των συζητήσεων. Ξέρετε ότι πιστεύω ότι πολύ καλή δικαστική συνεργασία θα πρέπει να εφαρμοστεί για την αποτελεσματική ε, ε αναγνώριση των αποφάσεων και για δίκες δίκες ε, θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις πολλές παραπομπές στο εθνικό δίκαιο από το κείμενο για να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εναρμόνιση και όσον αφορά τα δικαιώματα, το φυλάδιο με τα δικαιώματα που θα χορηγείται στον ύποπτο ε, δεν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις. Μετά τι άλλο έχει δρομολογηθεί. Η οδηγία για πρόσβαση, δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, σε νομικό, το ε, κολέγιο το σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υιοθετήσει αυτό το μέτρο τον Ιούνιο οπότε θα έχουμε ένα πραγματικό σύστημα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων. Αναφερόμενοι τώρα στα ατομικά δικαιώματα επεξεργαζόμενοι το θέμα των υπόπτων στις ποινικέ υποθέσεις κατάλαβα ότι τα θύματα δεν συμπεριλαμβανόταν πουθενά στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Γι' αυτό την περασμένη εβδομάδα υπέβαλα ένα πακέτο για τα δικαιώματα των θυμάτων που ασχολείται με την ποιότητα της προστασίας και της υποστήριξης στα θύματα μετά το έγκλημα και κατά τη διάρκεια των διαφόρων ποινικών διαδικασιών. Όλα τα θύματα έτσι θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας, υποστήριξης, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όποτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα ε, από πού κατάγονται, από ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάγονται ή πού διαμένουν. Τι είναι αυτό. Είναι μια νέα οδηγία, αυτό είναι αυτό το νέο πακέτο, που θεσπίζει σαφείς υποχρεώσεις, υποχρεωτικές υποχρεώσεις που πρέπει να συμμορφώνονται ε, τα κάτι με αυτές για την προστασία των θυμάτων και θα δίνεται στα θύματα η σωστή ε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεύτερο στοιχείο, ένας κανονισμός για την αμοιβαία αναγνώριση του, της προστασίας προβλέπει το αστικό δίκαιο και τα σχετικά μέτρα. Γιατί μόνο του αστικού δικαίου, διότι τα κράτη-μέλη αποφάσισαν αρχές του μήνα να περιορίσουν το πλαίσιο της πρότασής τους για την προστασία, τα μέτρα για την προστασία στα πλαίσια του ποινικού δικαίου, οπότε θα εφαρμόζεται αυτό αφού διαπραχθεί ένα έγκλημα και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολείται με το πλαίσιο του πολιτικού, ε, του αστικού δικαίου, τα προληπτικά μέτρα και αυτές οι δύο προτάσεις θα κινούνται μαζί για να δημιουργούν μια σφαιρική εικόνα που θα παρέχει ασφάλεια δικαίου για το θύμα ανεξάρτητα από τους εθνικούς κανόνες για την προστασία. Παντού η προστασία που θα παρέχεται θα είναι η ίδια παρόμοια, χωρίς διαφορές. Ε, είχα μια συζήτηση με τον πρόεδρό σας και γνωρίζω ότι οι πολιτικές ε, ομάδες γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποια θύματα που είναι πιο ευάλωτα από άλλα, είτε διότι υπάρχει κίνδυνος να είναι ξανά θύμα από, τον, ε, από αυτόν που διέπραξε το αδίκημα, είτε από τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά εντοπίζει και τις δύο κατηγορίες των ευάλωτων θυμάτων. Παιδιά, άτομα με αναπηρίες, θύματα σεξουαλικής βίας, θύματα εμπορίου ανθρώπων. Εντοπίζουμε και άλλους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατικών πράξεων, παραδείγματος χάρη, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα όσον αφορά τις απειλές και επανειλημμένες βιοπραγίες εναντίον τους. Οπότε ε, χρήζουν Ιδιαίτερη προστασία. Προτείναμε και τα μέλη τη οικογένειας των θυμάτων να έχουν τα ίδια δικαιώματα δυνάμει της οδηγίας όπως και τα άμεσα θύματα. Όχι μόνο τα άμεσα θύματα προστατεύονται, αλλά και οι έμεσα εμπλεκόμενοι που συνδέονται με τα θύματα θα προστατεύονται. Όπως μια μητέρα προστατεύει το παιδί της. Το παιδί είναι θύμα, η μάνα δεν είναι θύμα, αλλά αυτομάτω επειδή είναι θύμα το παιδί είναι και η μάνα θύμα. Πρέπει και οι δύο να προστατεύονται και η προτινόμενη οδηγία περιέχει πολλέ σημαντικέ προδιαγραφέ για δικαιώματα, υποστήριξη, προστασία, όλα αυτά που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θεωρώ αυτό ένα πρώτο βήμα σε μια συνεχή διαδικασία. Στο μέλλον θα πρέπει να αναλυφθούν περαιτέρω δράσεις, παραδείγματος χάρη για την αναθεώρηση των ισχυσών οδηγιών περί αποζημιώσεως θυμάτων εγκλημάτων θα αναλυθούν τα κενά υπάρχουν όσον αφορά την προστασία συγκεκριμένων κατηγοριών θυμάτων εγκλημάτων όπως τρομοκρατία οργανωμένο έγκλημα, βία βάση του φύλου. Σύντομη είναι αυτή η παρουσίαση κύριε Πρόεδρε, θα μπω σε λεπτομέρειε σύντομα διότι η Επιτροπή σας θα επεξεργαστεί αυτά τα θέματα, πιστεύω αυτό το πακέτο. Άρα θα επανέλθουμε σύντομα. Άλλο στοιχείο η μεταρρύθμιση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων. Καλωσορίζω το σχέδιο εκθέσεως του Άξελ Βος που λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και τονίζει πέντε σημαντικές πτυχές της, μετα... της μεταρρύθμισης, γενική προσέγγιση, ατομικά δικαιώματα, η διάσταση της εσωτερικής αγοράς, η επιβολή των κανόνων, και η γενική σφαιρική παγκόσμια διάσταση. Τώρα, η γενική ολιστική προσέγγιση. Περιμένετε πλήρη εναρμόνιση και ασφάλεια δικαίου που θα παρέχει ομοιόμορφη προστασία υψηλού επίπεδου των ατόμων σε όλες τις περιστάσεις. Αυτό ήταν παράθεση που έκανα τώρα και ε, αυτό είναι και ο δικός μου στόχος. Εναρμόνιση και ασφάλεια δικαίου. Απαιτούνται αυτά και για τους καταναλωτές και για τους οικονομικούς φορείς και σωστά υπογραμμίζεται ότι ο ίδιος βαθμός προστασίας των ατόμων χρειάζεται ανεξάρτητα από το που βρίσκεται εκείνος που ελέγχει τα στοιχεία. Αυτό θα περιέχεται στην πρότασή μου, διότι θα πρέπει να παρέχεται προστασία ανεξαρτήτως της τοποθεσίας του παρόχου των υπηρεσιών. Θεωρείται επίσης ότι ενα θεωρημενο καθεστώς προστασίας των δεδομένων πρέπει να μειώνει τη γραφειοκρατία και το διοικητικό άχθος, και εδώ συμφωνώ απόλυτα, θα πρέπει να περικοπεί η γραφειοκρατία και να εξαλειφθεί εξαλειφθούν διοικητικές υποχρεώσεις που δεν είναι αναγκαίες και είναι αναποτελεσματικές και να επικεντρώσουμε στα ελάχιστα, τις προσπάθειες στα ελάχιστα αναγκαία. Δεύτερο σημείο, τα ατομικά δικαιώματα. Εδώ μιλάμε για την έννοια της συνένεσης ε, τη συμφώνου γνώμη που είναι στο επίκεντρο. Θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων. Περί πρόκειται. Θα πρέπει να είναι ρητή η αναφορά. Και στην πρότασή μου τη σχετική θα αναφέρω χρειάζεται να είναι πολύ ξεκάθαρο. Ξεκάθαρη η, όροι συνθήκες. Η εσωτερική αγορά θέλετε να είναι υποχρεωτικός ο καθορισμός των υπευθύνων για την προστασία των δεδομένων. Εμείς δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ όσο το Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Δεν αποφασίσαμε κατά πόσο αυτή η αρμόδια προστασία των δεδομένων θα πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά ή όχι. Είμαστε εν το μέσο αξιολογήσεως. Θέλουμε να δούμε μέχρι πού θέλουμε να προχωρήσουμε από αυτού. Υπάρχει και άλλο συγκεκριμένο σημείο που υποστηρίζω πολύ, είναι η ενίσχυση και εναρμόνιση του καθεστώτος προστασίας των, των αρχών προστασίας των δεδομένων. Εδώ υπάρχει μια πραγματική ανάγκη, διότι αν θέλουμε οι κανόνες περί προστασίας των δεδομένων να λειτουργούν, τότε πρέπει να δώσουμε και ουσία, να δώσουμε ισχύ. 27 φορείς προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να είναι τα σαγόνια. Θέλω να δώσουμε δόντια λοιπόν στο, στους φορείς αυτούς. Όχι μόνο σαγόνια χωρίς δόντια. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω την καλύτερη δυνατή λύση. Τέταρτον, η γενική σφαιρική διάσταση της προστασίας των δεδομένων. Δίκιο έχετε, χρειάζεται εναρμόνιση των διαδικασιών, ενίσχυση για την μεταφορά διεθνών στοιχείων. Ε, να σας δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα. Να δημιουργήσουμε μηχανισμό ασφαλείας, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τρίτες χώρες, ασφαλείς λιμένες αποκαλούνται εδώ εισαγωγικών. Έχουμε ήδη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νέο στοιχείο θα είναι ο μηχανισμός υποχρεωτικός με εγγυήσεις για την εφαρμογή του, για τη λειτουργία του. Βλέπετε πολλά απομένουν να συζητηθούν. Απλώς ήθελα να σας δώσω μια πρώτη γεύση σχετικά με το που βρισκόμαστε όσον αφορά αυτά που μαγειρεύονται εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ελπίζω προς το τέλος του χρόνου να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο νομοθετικού κειμένου. Στις συνεχιζόμενες μας συζητήσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την προστασία των δεδομένων, εν ώψη συμφωνίας, ξέρω ότι η επικεφαλής των πραγματεύσεων, ο Γενικός Διευθυντής, η Διευθυντή, μάλλον Φρανσουάς Λεμπάι, ήδη σας έχει ενημερώσει σχετικά με τις ε, ε, διαπραγματεύσεις αυτές εχθές Τώρα, όσον αφορά την οδηγία περί ελεύθερης ε, διακίνησης και Σέγγεν, η δημιουργία μιας Ευρώπης άνευ συνόρων, όπου εκεί η ελεύθερη διακίνηση ατόμων εξασφαλίζεται, αυτό για μένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής ε, Ενώσεως και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο πρόεδρος Μπαρόσο επανειλημμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πρόθυμη να υποχωρήσει και να υπονομεύσει την ελεύθερη διακίνηση. Οι πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας έδειξαν ότι κάποιοι κανόνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως που αφορούν τη διακίνηση ατόμων που διασύνουν τα σύνορα πρέπει να ερμηνεύονται πολύ καλά και σωστά και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι οι εθνικές κυβερνήσεις δεν δίνανται να ορίσουν τους όρους και τις συνθήκες για την επανεισαγωγή ε, μεθοριακών ελέγχων μονομερός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν στεναρή όσον αφορά την ανακοίνωση της δανέζικης κυβερνήσεως που προτίθεται να εισαγάγει ενισχυμένους μεθοριακούς ελέγχους εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως βάζοντας μόνιμα τελωνιακούς ελέγχους στα δανέζικα σύνορα. Σε μια επιστολή τη 13 η Μαΐου, ίσως γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος Μπαρόσο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη συμβατότητα του μέτρου που εξετάζει ως ενδεχόμενο να εφαρμόσει η δανέζικη κυβέρνηση με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε προσωρινός μεθοριακός έλεγχος πριν αυτός εφαρμοστεί ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως περί ελεύθερης διακίνησης. Ιδιαίτερα τον κώδικα ε, για τα έλεγχο των συνόρων του Σέγγεν και γενικά το θέμα της ελεύθερης διακίνησης των ε, ατόμων. Το μήνυμά μας ήταν σαφέστατο. Ε, εμείς είμαστε στεναροί όσον αφορά τη θέση μας για τα δικαιώματα και τις αρχές που εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και βελτιώναμε την εφαρμογή της νομοθεσίας στην ελεύθερη διακίνηση, την οδηγία του 2004 για τα δικαιώματα των πολιτών και των μελών των οικογενειών τους να μετακινούνται και να διαμένουν ελεύθερα. Είχα διμερείς επαφές και με τα 27 κράτη-μέλη για να συζητήσουμε τα θέματα και να εντοπίσουμε πού βρίσκονται τα προβλήματα όσον αφορά την σωμάτιση οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Πάνω από τα μισά κράτη-μέλη έχουν ενσωματώσει, είναι καθοδόν ενσωμάτωση των κανόνων αυτών στη δική τους ένωμη τάξη, να εφαρμόσουν πλήρως αυτούς τους κανόνες. Άρα αυτό δείχνει ότι υπήρχαν προβλήματα πριν, Όσον αφορά τα ανεπίλητα προβλήματα με τα υπόλοιπα 12 κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει πλήρη εφαρμογή, ξεκινώντα και διαδικασίες κατά παράβαση όταν αυτό ενδείκνυται. Ε, παράλληλα, Έχουμε δώσει βοήθεια στα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τους κανόνες για ελεύθερη διακίνηση και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε αυτό όποτε χρειάζεται αυτό για να υπάρχει πλήρη συμβατότηση. Αυτό είναι σας δείξω ότι ακόμα και αν δεν ετοιμάζω συνέντευξη τύπου για αυτά τα θέματα κάθε δύο εβδομάδες, παρόλα αυτά γίνεται αυτή η δουλειά εκ των πραγμάτων. Διότι θέλω αυτή η οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση να λειτουργεί πλήρως και όχι μόνο εν μέρη όπως βρήκα να είναι η κατάσταση όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου ω Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για το εμπεδεσίωση του προγράμματος εργασία και τώρα να υπενθυμίσω πώς έχουν τα πράγματα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχουμε έναν κατάλογο, τουλάχιστον 20 μέλη θέλουν να πάρουν το λόγο και έχουμε πρόγραμμα λοιπόν, χρονικό όριο, ο γραμματέας Επιτροπής ε, Βενετίας ε, θα έρθει στις 11.30 εδώ, οπότε χρόνος ομιλίας δύο λεπτά προτείνω για καθέναν. Αλλιώ δεν θα έχουμε χρόνο. Δύο λεπτά στον κάθε βουλευτή. Δύο λεπτά μόνο παρακαλώ. για να μην συμπιέσουμε την υπόλοιπη ημερήσια διαταξή μας. Δύο λεπτά στον καθένα λοιπόν. Ξεκινάμε την κυρία Γιαρόκα. Δεν, δεν σας σημειώσα, αλλά αν θέλετε να πάρετε πρώτο το λόγο συντονιστής, παρακαλώ. Κύριε Μπουσούτιλ. Κύριε Μπουσούτιλ, ευχαριστώ την ε, Αντιπρόεδρο κυρία Ρέντινγκ Έχω μία ερώτηση και δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ερώτηση για το πακέτο θυμάτων και την ε, ε, σχέση της με το EPO. Ε, δεν καταλαβαίνω πώς αυτά τα δύο θα συγκλίνουν. Η πρόταση για το EPO θα καλύπτει την ε, ποινική πτυχή και η καινούρια σας πρόταση για κανονισμό θα καλύπτει την αστική πλευρά. Θα έχουμε δύο διαφορετικά νομοθετήματα που θα καλύπτουν τους ίδιους στόχους. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Μετά, προστασία των δεδομένων, παρατήρηση εδώ. Ε, Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε και χαίρομαι που λαμβάνετε υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου πριν υποβάλλετε πρόταση. Φαντάζομαι θα την υποβάλλετε τον Ιούλιο. Οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία την πρότασή σας για την αναθεώρηση οδηγίας προστασίας των δεδομένων. Και θα μιλήσουμε για αυτήν τον Ιούλιο. Μετά, για την ελευθερία κυκλοφορία των προσώπων. Μία ακόμα παρατήρηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 100% υπέρ σας για την προστασία της ε, Ευρώπης χωρίς σύνορα. Στην αρχή είχαμε ανησυχήσει. Φαινόταν η Κομισιόν να μην έχει σαφή άποψη. Αλλά καθώς περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες ε, αυτή η δισταγμή του οποίου εμεί θεωρούσαμε ότι είχε η Κομισιόν, μετατράπηκαν σε μια πραγματική θέληση προάσπισης της Ευρώπη χωρί σύνορα. Θέλω να το υπογραμμίσω γιατί είναι πολύ καλό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωρίζει ότι θα έχει σύμμαχό της το Κοινοβούλιο σε αυτόν τον αγώνα. Ευχαριστώ. Ωραία. Από τους σοσιαλιστές, η κυρία Φλασικό Βαμπένοβα. Όχι. Κυρία Γκάντς. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο ιδιαίτερα για την προάσπιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και ε, το κεκτημένο του Σέγγεν, την Ευρώπη χωρίς σύνορα. Ξέρω λοιπόν ότι ήρθατε σε είχατε διμερείς επαφές με, τις 27, με τα 27 κράτη-μέλη και ελέγχετε την κατάσταση σε όλα τα κράτη. Επίσης χαίρομαι για τη στρατηγική ένταξη στον Ρωμά και θα ήθελα να επαναλάβω και το εξής μας από ε, λίγο οι πτυχές κατά της διάκρισης αυτής της στρατηγικής του χρόνου όταν θα υποβάλλετε έκθεση για τα επιτεύγματα και τις αλλαγές ό,τι αφορά την ένταξη των Ρωμά σε όλες τις χώρες. Θα ήθελα να δώσετε μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την πτυχή, διότι σε μερικές ε, χώρες υπάρχουν παραστρατιωτικές ομάδες που δημιουργούν προβλήματα με τους πληθυσμούς Ρωμά και άλλες ομάδες και χρειάζεται να τις παρακολουθούμε πάρα πολύ κοντά, γιατί υπάρχει και η κοινωνική πτυχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ένφελτ. Ε, θα αποφύγω τις ευχαριστίες για όλα τα καλά που έχει κάνει η κυρία Ρέντινγκ, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Δύο ερωτήσει. Μία γενική καταρχήν. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ερμηνείας της χάρτας των θεμελιών δικαιωμάτων. Η Κομισιόν από ό,τι φαίνεται ερμηνεύει αυτή τη χάρτα συσταλτικά. Ότι δηλαδή εφαρμόζεται μόνο κατά την στιγμή που εφαρμόζεται η κοινωτική νομοθεσία. Στην πραγματική ζωή όμως τα κράτη-μέλη παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε μέρα. Είτε πρόκειται για δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, λεσβιών κλπ. Ελευθερίες έκφραση, ελευθερία τύπου, ελευθερία θρησκεύματος και ξεφεύγουν γιατί η Κομισιόν λέει «Α, αυτό είναι θέμα της επικουρικότητας» είχαμε ε, επιθέσεις σε δικαστήριο του Στρασβούργου για παράδειγμα που δεν είναι ευρωπαϊκό, θέμα ευρωπαϊκού δικαίου βέβαια αλλά θα ήθελα η Κομισιόν ε, να ακολουθήσει μια προσέγγιση όπως αυτή που ακολουθεί για τους κανόνες ανταγωνισμού ε, δηλαδή να είναι πολύ πιο πλατεί το πεδίο δράση τη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεύτερη παρατήρηση για τα δικαιώματα ομοφιλοφίλων, λεσβιών, ε, ε, και τραβεστή. Ε, αυτή η ομάδα χάνει τα δικαιώματά της μόλις περάσει τα σύνορα ε, ακόμα και την κυδαιμονία των παιδιών τους. Θα θέλαμε, έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν ένα οδικό χάρτη, όπως παρόμοιο με τον οδικό χάρτη της ισότητας των φύλων, και για αυτή την ομάδα. Η Κομισιόν ως τώρα δεν έχει προβεί σε τέτοιου είδους επεξεργασία ενός οδικού χάρτη. Θα ήθελα να το ξαναζητήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους πράσινους, κυρία Στέλοκα. Και εγώ θα αναφερθώ στο ίδιο θέμα για τις ε, ε, στενής ερμηνείας του άρθρου 51.1 της χάρτας, ε, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Ιντφέλτ. Η θέση των πρασίνων είναι ότι η Επίτροπος έχει υποχρέωση να αναλάβει δράση κατά κράτους μέλους όταν υπάρχει ζήτημα παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Θα θέλω να μας πείτε την άποψή σας. Δεύτερον, το έθιξα και όταν, συζητήσαμε, ε, όταν συναντήκαμε στο πλαίσιο των σκιωδών εισηγητών. Όταν αξιολογούμε την εφαρμογή της χάρτας όταν αξιολογείτε την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιών Δικαιωμάτων ε, δεν το κάνετε ανακράτος. Δεν αναφέρετε την επίδοση του κάθε κράτους σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, ίσως θα έπρεπε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Κομισιόν να αλλάξει αυτή την τακτική και ε, να κάνουμε αυτό που κάνουμε και με τις ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να αναφερόμαστε στην επίδοση του κάθε κράτους χωριστά και για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση. Γιατί να έχουμε αυτή τη διαφορά, τη διάκριση. Δεύτερον, για τα θέματα των ατομικών προσφυγών ενώπιον του ε, Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επί τη βάση της ε, χάρτας. Ποιο, ποια είναι η σκοπή σας, ποια είναι η στόχη σας σε ό,τι αφορά την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Ευχαριστώ για την ECR και ο Σκύρκοπ. Ευχαριστούμε την κυρία Ρέντινγκ. Δύο σχόλια έχω να κάνω. Χαίρομαι που τα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και η προστασία δεδομένων είναι προτεραιότητα. Περιμένουμε τις προτάσεις της. Συμμερίζομαι τις, ε, από, τις απόψεις για τους υποχρεωτικούς ε, υπεύθυνου ε, προστασίας δεδομένων. Όμως, θα, ε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί, όχι μόνο φιλόδοξοι, προκειμένου να καταφέρουμε κάτι πρακτικά. Δεύτερον, για το μηχανισμό αξιολόγηση της Schengen. Ελπίζω στη συζήτηση αυτή να έχουμε στο μυαλό μας ότι η αξιολόγηση δεν θα πρέπει να γίνει μόνο με τεχνικά μέσα, δεν θα πρέπει να ελέγχεται μόνο από κάμερες και από βάση δεδομένων. Θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι πάντοτε η αξιολόγηση είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή στην αξιολόγηση θα πρέπει να αξιολογούνται και οι άνθρωποι και το προσωπικό και η επίδοσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να αξιολογούμε ε, και τα αποτέλεσματα των δράσεων των ανθρώπων και όχι μόνο του τεχνικού εξοπλισμού. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ ο κύριο Σταβάρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε που είστε εδώ. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή της παρουσίασής σας. Ότι οι επιστολές που παίρνετε με παράπονα από πολίτες ε, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κατά δύο τρίτα συγκεκριμένα, ε, ξεφεύγουν από τις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Αυτό που ε, βγάζω εγώ, η δική μου ερμηνεία αυτού, είναι ότι ε, τα, οι πολίτες μας πιστεύουν ότι τα θεμελιώδη τους δικαιώματα βρίσκονται υπό πίεση και ε, στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα προασπίσει σε, όλες τις, σε όλα τα κράτη-μέλη. Συνεπώς, αντί να το δείτε αρνητικά ως άγνοια εκ μέρους των πολιτών μας για το τι είναι η επικορικότητα, θα πρέπει να το ερμηνεύσετε ως ένα ακόμα δείγμα ότι οι πολίτες μας στηρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στη δράση της ε, όταν βρίσκονται ενώπιον αδύναμων κρίκων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και η θέση της ε, ε Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον Ουγγρικό νόμο περί και το Ουγγρικό σύνταγμα ε, αποτέλεσε μια αδυναμία ε, ένα κενό στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για το πακέτο τα δικαιώματα των θυμάτων, ε, πολύ θετικά τα όσα είπατε. Ε, λαμβάνετε υπόψη την εκθέση Άλεξ Voss επίσης. Τέλος θα ήθελα να πω το εξής για τη Σέγγεν. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα τη χάνει σεβασμού η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και με την οδηγία μη διάκριση. Γιατί όταν μια χώρα αυξάνει τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, για παράδειγμα στα σύνορα μεταξύ Δανίας και Γερμανίας, αυτό δεν γίνεται για να δημιουργηθούν προβλήματα στην Δανέζικη μειονότητα που ε, μένει στο Σλέσβικ Χολστάιν για παράδειγμα. Ε, προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε ανθρώπους που είναι, ε, προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί να εμπίπτει στην οδηγία των, με μη διακρίσεων. Ο κύριος Μπρόνς. Ναι, μιλάτε για τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όμως σας υπενθυμάσω ότι υπάρχουν τρία κράτη-μέλη τα οποία έχουν αυτοαποκλειστεί από το χάρτη αυτών. Πλην όμως κάποιοι συνάδελφοι από την Επιτροπή των Σταγματικών Υποθέσεων μου λένε ότι μετά τη θέσπιση της Συνθήκης Λισαβόνας είναι άκυρη αυτή η αυτοαποκλεισμή και η τσεχική δημοκρατία από ό,τι φαίνεται... Ε, δέχθηκε να συνυπογράψει την συνθήκη της Λισαβόνας μόνο, μάλλον να κυρώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας μόνο μετά την εξασφάλιση ποτέ του αυτοαποκλεισμού, του opt-out. Άρα είναι θέμα εφαρμογής και εφαρμοσιμότητας ε, της χάρτας των θεμελιδών δικαιωμάτων για τα κράτη αυτά που έχουν αυτό αποκλειστεί ή όχι. Και όπως βλέπετε 30 δευτερόλεπτα μόνο χρειάστηκα. Ευχαριστώ πολύ η Επίτροπος τώρα για να δώσει τις απαντήσεις σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ κύριε Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που μου προσφέρατε και θα ήθελα εν συντομία να δώσω απαντήσεις σε κάποιες από τις ερωτήσεις. όσον αφορά τον, ε, την εντολή προστασίας. Ε, τα κράτη-μέλη, από ό,τι γνωρίζω, έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, να περιορίσουν το πεδίο της πρότασής τους ως προς την, ε, τις διαδικασίες προστασίας ποινικού δικαίου. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν συμπεριέλαβα στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων πρόταση ε, δεν έθεσα μάλλον προς πρόταση για την προστασία αυτή, γιατί υπάρχει αυτή η πρόταση των κρατών μελών. Έχω θέσει μόνο μία πρόταση για, το, για τα μέτρα του ποινικού δικαίου, του αστικού δικαίου, συγγνώμη, και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δουλέψουν μαζί. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ενδιάμεση διαδικασία, θα υπάρχει άμεση εφαρμογή ανεξαρτήτως του τι ορίζει το δίκαιο σε κάθε κράτος μέλος. Μία πρόταση δηλαδή των κρατών μελών θα περιορίζεται στο ποινικό δίκαιο, ενώ η πρόταση της Επιτροπής θα περιορίζεται στο αστικό, με, κάποιες, ε, με κάποια γεφυρώματα, με κάποιους συνδέσμους ως προς τις προτάσεις των κρατών μελών ώστε να γίνει απρόσκοπτα η μετάβαση. Αν και πρέπει να επισημάνω ότι θα πρέπει να είχαμε ήδη αυτό το, αυτή τη δυνατότητα συνεργασία. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Αλλά, πάση περιπτώσει. Προστασία των προσωπικων δεδομένων Ιούνιο-Ιούλιο. Αποφάσισα να το καθυστερήσω λίγο. Γιατί μπορεί να υπάρχει συμπληρωματική αξιολόγηση από τις διάφορες ε, προτάσεις που έχω δεχθεί και γιατί θέλω αυτό που θα σας προτείνω τελικά να είναι και νομικά στέρεο. Δεν θα αφορά δηλαδή μόνο την ε, επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον έξω κόσμο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζήτησα και μια δεύτερη μελέτη αξιολόγησης. Γι' αυτό θα καθυστερήσουμε. Δεν θα προλάβουμε πριν τις τερινέ διακοπές να καταθέσουμε την πρόταση. Ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή τόσο μέσω του Προέδρου, όσο και μέσω της κυρίας Μάλστρομ, όσο και της υποφαινομένης, έχει καταστήσει πιστεύω απόλυτα σαφές ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με η αδίποτε αρχή της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας. Δεν θα δεχθούμε η αδίποτε ή οδήποτε υποβιβασμό του, του κεκτημένου του Σέγγεν. Θα θεσπιστεί ο κώδικας Σέγγεν όπως πρέπει και όταν πρόκειται να γίνει, όταν γίνει αξιολόγηση που βέβαια δεν μπορεί να έχει σαν συνέπεια ότι θα υποβιβαστεί ο κώδικα Σέγγεν, απλώς θα εξηγεί αυτή κάποιες ερωτη... κάποια ζητήματα, θα δίνει απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Ε, ελεύθερη κυκλοφορία επίσης. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές, από τις βασικές αρχές και γι' αυτό και όταν εξέτασα την οδηγία περί ελεύθερης κυκλοφορίας του 2004 και τον τρόπο με τον οποίο αυτή είχε ε, μεταφερθεί, είχε εφαρμοστεί, ε, ξεπλάγιν, διότι ήταν ε, η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία πολύ ελλειπής. Και αυτή τη δουλειά ξεκίνησα, την ξεκίνησα από πέρσι την Άνοιξη, με αποτέλεσμα αυτό που σας περιέγραψα νωρίτερα, ότι τώρα πια έχουμε φτάσει σε ένα καλό στάδιο που μας επιτρέπει πιστεύω σύντομα να μπορούμε να πούμε ότι έχουν όλοι ευθυγραμμιστεί και εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες. Και τα δικονομικά δικαιώματα επίσης που προκύπτουν, που απορρέουν από την οδηγία για την ελεύθερη ε, κυκλοφορία, που είναι δικονομικά δικαιώματα του ιδιώτη, του ατόμου. Τώρα και αυτά έχουν ενσωματωθεί στο μέγιστο βαθμό στους εθνικούς κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, όπου ε, εκεί πραγματικά είχαμε τις μεγαλύτερες ελλείψεις. Και εκεί ακριβώς και το ζήτημα των Ρωμά ετέθη με μεγάλη έμφαση. Εκεί ακριβώ εντοπίζεται το μεγάλο μέρο των δυσκολιών σχέση με του Ρωμά, γιατί δεν είχαν διασφαλιστεί τα δικονομικά του δικαιώματα. Αυτά λοιπόν. Δεν υπάρχει κανένα συμβασμό στην υπόθεση αυτή. Δεν δεχόμαστε κανένα συμβασμό. Για του Ρωμά και τι διακρίσει. Ναι, γιατί υπάρχει διακρίση. Να σα πω απλούστατα, διότι υπάρχουν οι οδηγίε και εφαρμόζονται και όπως είπα ε, χρειάστηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές για την οδηγία περιελεύθερη κυκλοφορίας ώστε να ενσωματωθούν, να εξασφαλιστούν τα δικονομικά δικαιώματα. Έχουμε την οδηγία RACE και εάν τα πράγματα δεν δουλεύουν, ε, δεν προχωρούν όπως πρέπει, θα χρειαστεί να καταφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με διαδικασίες παραβιάση, όπως άλλωστε κάνω τακτικά και συστηματικά και το γνωρίζουν τα κράτη-μέλη πολύ καλά, ότι όταν δεν πάνε τα πράγματα όπως όφυλαν, όταν δεν κάνουν αυτό που όφυλαν τα κράτη-μέλη, σε μια περίπτωση μεταφοράς εθνικών δίκαιο ε, οδηγίας, επικρέμεται η διαδικασία επί Τώρα, γιατί ειδικά ένα πλαίσιο για τους Ρωμά, για τις στρατηγικές Ρωμά, κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία. Γιατί τα εντάξαμε, γι' αυτά υπογραμμίσαμε αυτό ιδιαίτερα. Γιατί είναι όρια εκ των όνων κάνευ για την ενσωμάτωση. Εάν τα παιδιά τους δεν πάνε σχολεία και μόνο 32% των παιδιών των Ρωμά, σε σχέση με 97% των παιδιών του γενικού κοινού θα έλεγα, ε, δεν πάνε, ε, είναι μόνο αυτά τα οποία πάνε στο δημοτικό. Εάν δεν πάνε στο δημοτικό λοιπόν μετά πάλι θα είναι θέματα ε, διακρίσεων. Εάν δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στι υγειονομικέ υπηρεσίε, στι υπηρεσίε υγεία και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε και τα παιδιά, προφανώς δεν μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω στη ζωή τους. Αυτά είναι και ο λόγος για τον οποίο ζητώ από τα κράτη-μέλη σαφείς προτάσεις για το πώς σκοπεύουν να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό μέχρι τα τέλη του έτους και Περιμένω τις, από, τις προτάσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτάσουν μέχρι τα τέλη του έτους. Φυσικά θέλει διαφορετικές ανακράτως μέλος γιατί και τα πληθυσμιακά στοιχεία στο κάθε κράτο μέλο είναι διαφορετικά. Κάθε κράτο μέλο έχει διαφορετική κατάσταση. Κάθε κράτο μέλο, όπω και το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, θα πρέπει να καταθέσουν προτάσεις. Είναι κοινή ευθύνη σε μια διαφορετική σε ανάληψη διαφορετική δράση, μεν ανάλογα με τα προβλήματα που έχει ο καθένα, αλλά μετρήσιμη δράση. Και γι' αυτό ακριβώ οι προτάσεις θα κατατεθούν και θα επαληθευθούν και έχω στήσει και από την υπηρεσία της Βιέννης να μας δώσει στοιχεία σε συνεργασία και με το Συμβούλιο της Ευρώπης να προχωρήσει αυτή η παρακολούθηση της υλοποίησης ώστε να δούμε πώς η πρόοδος σημειώνεται, πού εντοπίζονται τα κενά. 26,5 δις ευρώ είναι διαθέσιμα και ενδεχομένω θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Πώς λοιπόν μπορούν να φτάσουν τα χρήματα αυτά στους δικαιούχους χωρίς να χαθούν μέσα σε project τα οποία δεν έχουν απτέ λύσεις να προσφέρουν. Όλη αυτή η διαδικασία της παρακολούθηση. ή ο έλεγχος από του ε, από τους εταίρους, το peer review, Όλα αυτά είναι μέσα στις προτάσεις μας και θα επανερχόμαστε κάθε χρόνο για να, ε, ενώπιον του Κοινοβουλίου για να σας εξηγούμε πόσο έχουμε προχωρήσει και πού φτάνουμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα όπως άλλωστε χρειάζεται. και βλέπω εδώ την κυρία Λίβια Ζωόκα, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε τεράστια σημασία, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ένωσαν τη φωνή τους για να πούνε πρέπει να γίνει κάτι. Δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε όλα τα κράτη-μέλη. Πολλά ήταν πολύ διστακτικά. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω τώρα για, την, ε, για τα καλά νέα ότι όντως τώρα τους έχουμε κερδίσει όλους, συμπράττουν όλοι. Θα πρέπει να πω ότι ένα μικρό θαύμα έγινε και μπορέσαμε να κερδίσουμε τα κράτη-μέλη, τα βοηθήσατε κι εσείς να βγουν από αυτή την αρνητική στάση και να ακολουθήσουν όλα τον ίδιο δρόμο πια, τον ίδιο στόχο. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο δεν βγαίνει από την ημερήσια διάταξη, αντίθετος είναι πάντα επικαιρότητα. Τώρα η χάρτα, γιατί είναι ε, στενή ερμηνεία. Εγώ δεν βλέπω πουθενά στενή ερμηνεία. Πρόκειται απλώ για το άρθρο 51. Δεν έβαλα εγώ το άρθρο 51 στην χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη το έθεσαν, το συμπεριέλαβαν γιατί δεν ήθελαν να έχουν συνέχεια στο σβέρκο του, στο χρόνο τη Επιτροπή. Η Επιτροπή ω θεματοφύλακα συνθήκη είναι υποχρεωμένη να επαγρυπνεί για την τήρηση συνθήκη. Εάν δεν σα αρέσει το άρθρο 51, διαγράψτε το. Εξασφαλίστε την απάλληψή του υπό τη συνθήκη. Όσο όμω ισχύει το άρθρο 51, το οποίο ξεκάθαρα λέει ότι όπου έχει, ε, ορίζει μάλλον που έχει εφαρμογή και που δεν έχει εφαρμογή ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εμεί δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πράξουμε και έχω αρχίσει πολύ συγκεκριμένα να το διατυπώνω στο εγχειρίδιο το οποίο συντάσσουμε ε, για τον εορτασμό του πρώτου έτους εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπου έχουμε καταγράψει όλες τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα των πολιτών για να επισημάνουμε συγκεκριμένα πού εντοπίζονται τα προβλήματα, σε ποιο βαθμό και πώς πρέπει να προχωρήσουμε για να εξασφαλίσουμε την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Το πού θα γίνει αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να γίνει αυτή η δουλειά. Έτσι λοιπόν ε, το σεμινάριο που σκοπεύουμε να έχουμε τον Οκτώβριο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Επιτροπή των Αναφορών, η δική σα. οι Επιτροπές Αναφορών των Εθνικών Κοινοβουλίων, οι διαμεσολαβητές, ο, εθνικός, ο Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής και η Εθνική. οι εθνικοί οργανισμοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα έχουν αποτελέσει ένα ευρύτατο πεδίο ανα, ε, ανάλυσης μελέτης αυτής της κατάστασης, των προβλημάτων, των απαντήσεων που πρέπει να δίνονται σε παραβιάσεις δικαιωμάτων και αν δεν δίνονται σωστές απαντήσεις τότε θα πρέπει κάτι να αλλάξει, τε πρόκειται για το ευρωπαϊκό επίπεδο και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όπως ξέρετε και εγώ έχω από πλευρά μου εισαγάγει τον ε, κατάλογο επαλήθευσης θεμελιωδών δικαιωμάτων, Human Rights, ε, Fundamental Rights Checklist ε, και βλέπω ότι και τα κράτη-μέλη τον χρησιμοποιούν για να επαληθεύουν ότι όντως τηρούνται όπως οφείλουν τα κράτη-μέλη και ελπίζω να κάνει και το, και το Κοινοβούλιο την ίδια δουλειά ώστε και τα τρία θεσμικά όργανα να έχουν αντίστοιχη προσέγγιση στο θέμα. Οι εθνικές θεσμικές, τα εθνικά συντάγματα, το Δικαστήριο του Στρασβούργου Ξέρετε ότι έχουν τον ίδιο στόχο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι έχουμε και ένα ζήτημα για την έγκριση της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου, μάλλον την προσχώρηση της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και πιστεύω ότι μετά τον Αύγουστο θα είμαι σε θέση να σας ε, ε, πληροφορήσω για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να κλείσει και το θέμα αυτό και να υπάρχει επαλήθευση διπλή πλέον, όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων το οποίο πάλι θα κρίνει δυνάμει του χάρτη. Καινούριο στοιχείο. Είχα την πρώτη Είχα μια συζήτηση πριν από λίγο καιρό με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, το οποίο πλέον θα μπορεί να κρίνει με βάση το χάρτο θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, προσωπικές ατομικές ε, δηλαδή προσφυγές και είναι πολύ μεγάλη η ικανοποίηση που μας δίνεται από το γεγονός ότι και τα δύο δικαστήρια του Λουξεμβούργου, δηλαδή και του Στρασβούργου, το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους για μια κοινή αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων, δηλαδή ώστε ε, να χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο αυτές τις υποθέσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να μην μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου και να μην έχουν ούτε αντιφατικές αλλά ούτε επικαλυπτόμενες αποφάσεις. Αυτή είναι μια πραγματικά επικοδομητική συνεργασία. Ένας πολίτη μπορεί να προσφύγει σε εθνικό δικαστήριο, εάν τη ζήτημα ευρωπαϊκού δικαίου, το εθνικό δικαστήριο παραπέμπει για προδικαστικό ε, ζήτημα το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και από εκεί παίρνει μια προδικαστική απόφαση. Οι δε υποθέσει οι οποίε έχουν φτάσει ή μάλλον κατατίθενται πλέον για κρίση στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου έχουν ραγδαία ανάπτυξη και ακόμη δεν έχουμε αρχίσει καν, δεν έχουμε αντιληφθεί καν τι δυνατότητε του προσφέρει αυτή η νέα συνθήκη. Ε, και άπαξ και το αντιληφθούν και νομίζω ότι στην Επιτροπή των Σταγματικών Υποθέσεων έχουμε το θέμα αυτό τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου γιατί θα έχει τεράστιο φόρτο εργασίας, τεράστιο αριθμό υποθέσεων με τις, με τις ατομικές προσφυγές που θα ε, κατατίθενται πλέον. Άρα πλέον δεν μένει ακάλυπτος τομέα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μένει κενό, δεν μένει παράθυρο ανοιχτό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε ένα ε, πεδίο πλήρους καλύψης των ανθρώπινων δικαιωμάτων με απρόσκοπτη μετάβαση από την εθνική στην ευρωπαϊκή διάσταση για την προστασία των ατόμων. Επίσης, Ξέρετε, για το θέμα των ε, ομοφιλοφίλων ε, φιλομεταβατικών, ε, ξέρετε ότι έχουμε τακτικά επαφή με τους εκπροσώπους τους. Είχαν μάλιστα μία έκθεση στο κτίριο της Επιτροπής. Μάλλον τα έχουμε, έχουμε γίνει πολύ προοδευτικοί τελευταία. Έγινε λοιπόν η σχετική έκθεση. Ε, δεν ε, υπήρξαν αντιδράσεις δυσμενείς. Ο κόσμος έδειξε ενδιαφέρον, παρακολούθησε τα εκθέματα, ε, έθεσε και σε ερωτήσεις του. Άκουσα και εγώ τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες των εκπροσώπων ε, των ε, μοφιλοφίλων, ε, λεσβιών, φιλομεταβατικών. Πολλές φορές ακούσαμε και προσωπικές ιστορίες, μαρτυρίες. Είμαι λοιπόν ενήμερη για το θέμα αυτό, τα δικαιώματά τους και τα κενά στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. προστασία προσωπικών δεδομένων. Έχω δώσει νομίζω απαντήσεις στα περισσότερα από τα ερωτήματα. Σημειώνω επίσης και πάνω απ' όλα ότι έχουμε ένα ακόμη χρονικό περιθώριο μερικών μηνών για την κατάθεση των προτάσεων. Έχουμε ήδη λάβει υπόψη όσα έχετε προτείνει εσείς. Για ορισμένα έχει κλείσει το θέμα, για κάποια άλλα ακόμα θέλω να τα μελετήσω για να καταλήξω στις θέσεις μου. Πάντως, οι κανόνες οι οποίοι τίθενται προς ε, ε, λήψη αποφάσεων θέλουμε να είναι απόλυτα στέρεοι νομικά, να μην υπάρχει κανένα κίνδυνο να ανατραπούν, για να εξασφαλίσετε και η σχετική ασφάλεια δικαίου. Οι δε αρχές εθνικές ή ευρωπαϊκές προσφέρειες των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι ισχυρές, να έχουν ε, δόντια κοφτερά όπως λέμε, να ισχύουν για τους πάντε και να επιφέρουν τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης. Η προστασία δηλαδή του ατόμου είναι ξεκάθαρο ότι επεκτείνεται μέχρι και, την, μέχρι και τον τομέα των νέων τεχνολογιών. Όλα αυτά είναι σαφές ότι θα καλυφθούν από την νομοθεσία. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much for the answers. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, απαντήσεις. Έχουμε άλλα 13 μέρη που θα να υποβάλουν ερωτήσεις και έχουν κάποια σχόλια. Λοιπόν, θα έρθει μετά η Επιτροπή της Βενετίας. Έχουμε, μείνει, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας κατά μερικά λεπτά. Παρακαλώ ένα λεπτό καθένας για να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Äh, äh, λοιπόν, σας παρακαλώ ένα λεπτό για κάθε παρέμβαση για να τα βγάλουμε πέρα. Η ε, κυρία Γιαρόκα, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Το κοινοβούλιο σας είναι ευγνώμων Καθίστατε δυνατό το θαύμα με στο προσπαθειών σας. Όταν έθεσα τα ερωτήματα της Ρωμά, απαντήσατε σε όλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε ε, πολύ στεναροί όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Και το ερώτημά μου είναι το εξιστό. Από τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ετοιμάσουν τα εθνικά σχέδια δράση. Οι ομάδε δράση ή task force εργάζονται ω φορέα διευκόλυνση ή οι task forces εργάζονται ως φορέα διευκόλυνση ή task force μάλλον. Ε, υπάρχουν πολλές, ε, θα υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις μαζί σας τα κράτη-μέλη για να συνεργαστούν στο μέλλον και μας ρωτούν τι στρατηγικές πρέπει να ετοιμάζουν τα κράτη-μέλη. Ποιες είναι οι βασικές κατευθυντικές γραμμές που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορούν τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν ότι θα περάσει η στρατηγική τους ε, το Δεκέμβριο του 2011. Ποια είναι η απόψή σας. Ίσως καλό θα ήταν να συζητηθεί από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συζητείτε αυτό. Πώ μπορούν να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν. Ε, η κυρία Φλότρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ ήθελα να επανέλθω στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ένταξη των Ρώμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει μια στρατηγική για οικονομικούς πόρους. Θα δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη όταν ετοιμάζονται εθνικά σχέδια δράσης διότι η ποιότητα των σχεδίων θα εξαρτάται από τον τρόπο κατάρτισή τους. Τι θα ληφθεί υπόψη στα εθνικά σχέδια Εκεί η Task Force μπορεί να παίξει ένα ρόλο απέναντι στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Έτσι υπάρχει εγγύηση ότι υπάρχει συμμετοχή τοπική τοπικής αυτοδιοίκησης ενώσεων κοινωνικών εταίρων στην επεξεργασία των στρατηγικών. Και κάτι άλλο που θεωρώ ότι είναι αδύναμο στρατηγική. Η πρέπει, επαγρύπνηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία και κατά των διακρίσεων. Με τα χαράς βλέπω ότι δίνεται μεγάλη προσοχή στο θέμα. Βλέπουμε έναντι των Ρώμα να στρέφεται η γραφειοκρατία ε, των κρατών μελών, του δημιουργεί εμπόδια στη Γαλλία. Ναι, Κατάχρηση της, του δικαιώματος διαμονής. χρησιμοποιείται ένα ψευδές σχέδιο εθελοντικής επιστροφής των Ρώμα απέναντί τους. Και τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται είναι τεράστια εμπόδια για το να επιτρέψουν στους Ρώμα από τη Βουλγαρία και την Ρωμανία να ενταχθούν σε μια βιώσιμη στρατηγική. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, ε, να μείνετε στο ένα λεπτό. Ο κ. Παπα-Νικολάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είσαστε μαζί μας για άλλη μια φορά. Είπατε στην αρχή της παρουσίασή σας ότι υπάρχει η πρώτη, προ... η πρώτη έκθεση προόδου για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που αποδειγμένως ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, συνήγος του πολίτη, έκανε μια ε, έρευνα. 72% των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με αυτή, πιστεύουν ότι δεν ενημερώνονται επαρκώ όσον αφορά τα δικαιώματά τους που διαφυλάσσονται από την χάρτα, προστατεύονται τη χάρτα, 7% δεν γνωρίζουν καθόλου ότι υπάρχει χάρτα, 42% από αυτούς που συμμετείχαν είπαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διαφάνεια ε, που επικρατεί στην ευρωπαϊκή διοίκηση. Έχετε κάποια σχέδια για το μέλλον, για να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών να γνωρίζουν καλύτερα οι Ευρωπαίοι πολίτες τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη χάρτα. Ευχαριστώ. Έμαθα, λέει η Πρόεδρος, ότι η κυρία Επίτροπος πρέπει να φύγει. Δεν μπορούμε να θέσουμε όλα τα ερωτήματά σας. Θα πάμε στις γραπτές ερωτήσεις. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ισορροπία μεταξύ ομάδων. Θα ζητήσω από την κυρία Λούτφορντ την κυρία Λάτφορντ να υποβάλει ένα ερώτημα και μετά θα σταματήσουν οι προφορικές ερωτήσεις και θα ζητήσουν την κυρία Επίτροπο να απαντήσει εν συντομία και ελπίζω να έχουμε την τύχη να σας ξανασυναντήσουμε και να υποβάλουμε γραπτός ενδεχομένως τις ε, υπόλοιπες ερωτήσεις. κυρία Λάτφορντ, σας είμαι ευγνώμων, λυπούμε τους άλλους όμως. Πέντε λεπτά να πω σας παρακαλώ οι συντονιστές να εξετάσουν το θέμα πώς ρυθμίζουμε αυτές τις ε, συνεδριάσεις. Εντάξει, και σέβομαι το χρονοδιάγραμμα της Επιτρόπου. Έχω δύο ερωτήσει. Το πρώτο, πιστεύω ότι η χάρτα, οι περιορισμοί της χάρτας πρέπει να τηρηθούν, οι νομικοί περιορισμοί σχετικά με το σε, σε ποια πράγματα εφαρμόζεται η χάρτα, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν. Ε, τα κατημελέχουμε το άρθρο όμως 6-7 στη συνθήκη που δίνει μια πολύ ευρύτερη βάση για ε, πολιτικές πρωτοβουλίες. Επί ευρέως φάσματος θεμάτων που άπτονται δημοκρατίας κράτου δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν σπρώχνει και τα όρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την απόψη μου. Δεύτερον, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, φαίνεται να υπάρχει σειρά αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δημιουργούν σύγχυση. και φαίνεται να υπάρχει προβλήματα όσον αφορά τα δικαιώματα που από τη θαγένεια κάτω μέσω τη ε, Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και δικαιωμάτων που απορρέουν τη χάρτα και ότι υπάρχει διαφοροποίηση δικαιωμάτων όταν μετακινείται κάποιος από ένα μέλος και πάει σε άλλο κάτω μέλος και όλα αυτά δημιουργούν πραγματικές ε, αντιφάσεις. Yes. The point is that... Υπάρχει ακόμα ένας κατάλογος μελών που ε, επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις, αλλά η Επίτροπο Ριστικός πρέπει να φύγει, οπότε προτείνω να χρησιμοποιήσουμε τη γραπτή διαδικασία. Θα ενημερώσουμε γραπτό την ε, Επίτροπο, θα της υποβάλουμε τις γραπτές ερωτήσεις και θα δώσει και η ίδια γραπτός απαντήσεις. Τώρα θα της δώσω το λόγο να απαντήσει σε ερωτήσεις που έγιναν ήδη. Ευχαριστώ. Έτσι είχε προβλεφθεί. Είχαμε προβλέψει μία ώρα για αυτή τη συζήτηση. Ε, έχω προγραμματίσει και εγώ μία ώρα στην ατζέντα μου και έχω κανονίσει να επισκεφθώ και άλλες επιτροπές. Λυπάμαι πολύ. Να επιστρέψω πάντως, αν, θεωρείτε, αν το θεωρείτε απαραίτητο. Πρώτον, για το θέμα της χάρτας. Σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες, από όλα τα κράτη-μέλη. Είχαμε συζητήσει την εφαρμογή του, της χάρτας εδώ στο Κοινοβούλιο ε, με παρουσία ελάχιστων μελών του Κοινοβουλίου. Ελάχιστον. Ίσως το φθινόπωρο θα έπρεπε να ξαναδιοργανωθεί μια συνάντηση που θα συζητήσουμε πάλι με τους εμπειρογνώμονες και του δικαστηρίου ε, το θέμα της ε, εφαρμογής της χάρτας. Το θέμα ε, των εθνικών στρατηγικών για τους Ρωμά. Νομίζω θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της η Task Force για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην επεξεργασία των εθνικών τους πολιτικών. Στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε τα κράτη-μέλη λέγοντας η στρατηγική σας δεν είναι καλή. Αυτό που επιθυμούμε είναι να ε, σχεδιαστούν οι καλύτερες πρακτικές και μετά θα δούμε και το πώς εφαρμόζονται. Εκεί μπορεί να γίνουμε πιο επικριτικοί. Και θα εξετάσουμε βέβαια και τις, ε, τη, τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα. Η Task Force ε, είπε ότι είναι διαθέσιμα 26 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διάφορα ταμεία και τις διάφορες ε, ε πολιτικές. Οπότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουν τους πληθυσμούς Ρωμά. Ε, θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την πολιτική καταπολέμηση της φτώχειας των Ρωμά. Στη στρατηγική 2020 βλέπουμε τη φτώχεια και την παιδεία ως ε, βασικούς πυλώνες. Συνεπώς, για αυτούς τους ευάλωτους πληθυσμούς, μεταξύ των οποίων είναι και η Ρωμά βέβαια, ε, θα πρέπει να ακολουθηθούν και αυτοί οι δρόμοι. Εμείς ε, θέτουμε στη διάθεση των κρατών μελών τεχνική συνδρομή, έτσι ώστε να αποκτήσουν πιο εύκολα πρόσβαση σε κονδύλια ταμείων και πολιτικών, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν εκμεταλλεύονται τα κράτη-μέλη. Είναι αλήθεια επίσης ότι οι, περισσότερα, οι περισσότεροι συμπολίτες μας δεν είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, ούτε σε, για το ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε για το εθνικό επίπεδο. Έχω λάβει ε, υποθέσεις, επιστολές για υποθέσεις διαζυγίων από ανθρώπους που ελπίζουν ότι μπορώ εγώ να τους βοηθήσω, δεν γνωρίζουν σε ποιον να απευθυνθούν εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε να ενημερώσουμε, να ενημερώνουμε. Αλλά πάντοτε ένα ψηλό ποσοστό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάλι δεν θα γνωρίζουν. Οπότε ναι στην ενημέρωση, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται να έχουμε και ένα δίκτυο που θα επιτρέπει αυτός ο οποίος παίρνει ε, ένα παράπονο, μια επιστολή και δεν είναι αρμόδιος να μπορεί να το προωθεί στον αρμόδιο υπεύθυνο. Αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Όταν ήμουν ε, πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, 30 χρόνια πριν, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχα συνδέσει τις Εθνικές Επιτροπές ε, Αναφορών των Εθνικών Κοινοβουλίων με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή προκειμένου ακριβώς να διοχετεύσω αυτές τις ε, αναφορές που ερχόντουσαν στο Κοινοβούλιο και για τις οποίες δεν ήταν αρμόδιο το Κοινοβούλιο στις Εθνικές Επιτροπές και στον ε, Διαμεσολαβητή. Ακριβώς για να βρει κάθε μία τη θέση που της αντιστοιχεί. Συνεπώς ναι στην πληροφόρηση, αλλά ταυτόχρονα και ένα δίκτυο αρμοδίων υπευθύνων για να απαντήσουν σε αυτές τις αναφορές. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Και πάλι λυπάμαι που δεν είχαμε αρκετό χρόνο να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά θα απαντηθούν γραπτός από την Επίτροπο Reading και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συνεχιστεί η συζήτηση για το πρόγραμμα εργασίας 2011-2012. Είμαστε έτοιμοι για τον Γενικό Γραμματέα της ε, Επιτροπής Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε δύο λεπτά θα έρθει.

Colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή αργούμε, σας παρακαλώ να ξαναρχίσουμε με το σημείο 21 στάδιο εκπόνηση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Βενετίας σχετικά με το Σύνταγμα της Ουγγαρία, όπως εγκρίθηκε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο στις 18 Απριλίου 2011. Η γνωμοδότηση προβλέπεται να εγκριθεί στις 17-18 Ιουνίου από την Επιτροπή της Βενετίας. Παρόν εδώ, ο γραμματέας της Επιτροπής της Βενετίας συμβουλευτικού οργάνου για, το, για την εφαρμογή του, των δικαιωμάτων του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη με βάση τις προδιαγραφές που έχει προσδιορίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλο μάλλον ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων και καλωσορίζω τον κύριο Τόμας Μάρκερ. Θα ακούσουμε την παρουσίασή του Επιτρέψτε μου μόνο να υπενθυμίσω ότι το Μάρτιο του 2011 κατόπιν αιτήματος ε, του Ουγγρικού Κοινοβουλίου η Επιτροπή της Βενετίας υιοθέτησε μια γνωμοδότηση για τη διαδικασία αυτή στην οποία Ξέφρασε ανησυχίες για κάποιες πτυχές τόσο της διαδικασίας όσο και του ουσίας αυτής της ε, αναθεώρησης. Και τώρα ετοιμάζεται η γνωμοδότηση που θα υιοθετηθεί στις 17 και 18 Ιουνίου, σε μερικέ εβδομάδες δηλαδή. Θα ακούσουμε λοιπόν την, παρακολούθη, την ε, παρουσίαση για το στάδιο εκπόδυνσης αυτής της γνωμοδότησης Παρακαλώ κύριε Μάρκετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που με καλέσατε ενώπιον της Επιτροπής σας. Πριν μπω στην ουσία του θέματος, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την Επιτροπή της Βενετίας, γιατί ίσως να μην τη γνωρίζετε τόσο καλά όλοι. Η Επιτροπή της Βενετίας είναι ένα συμβουλευτικό σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα συνταγματικά απαρτίζεται από ανεξάρτητους ειδικού που διορίζουν οι κυβερνήσεις, κυρίως καθηγητές του δημοσίου, δικαίου ή ε, ανώτατοι δικαστές ε, από σταγματικά δικαστήρια ή ανωτατα δικαστήρια. Σημαντικό για σας είναι ότι το, η Επιτροπή της Βενετίας δεν κάνει μελέτες για κάποιες χώρες μόνο ε, με δική του πρωτοβουλία, αλλά μόνο κατόπιν αιτήματο των κρατών μελών, των ίδιων των κρατών δηλαδή. Στην περίπτωση τη Ουγγαρία, μας ζήτησε το Ουγγρικό Κοινοβούλιο καταρχά, να μελετήσουμε τρία συγκεκριμένα και τεχνικά ζητήματα για το στάδιο αυτό τη προετοιμασία δραματικής μεταρρύθμισης και τώρα η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη μα έχει ζητήσει να εξετάσουμε το κείμενο της, ε, του συντάγματος στο σύνολό του. Άρα αυτή η γνωμοδότηση για τις τρεις ερωτήσεις που, ε, που είχαν υποβληθεί από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας έχει ήδη ετοιμαστεί και μπορώ να δώσω απαντήσει. Η άλλη δεν θα υιοθετηθεί αυτή δηλαδή που προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Θα εγκριθεί 17 και 18 Ιουνίου και ω εκ τούτου δεν έχω ακόμη έτοιμο το κείμενο. Το κείμενο θα είναι διαθέσιμο μόνο μετά την έγκριση του και ω εκ τούτου ε, προ το παρόν δεν μπορώ να σα δώσω πλήρη επισκόπηση για το έργο αυτό τη Επιτροπή τη Βενετία. Μόνο ορισμένα θέματα που θα μας απασχολήσουν στην γνωμοδότησή μας για το δεύτερο αυτό θέμα, όπως σας είπα. Για την πρώτη όμως γνωμοδότηση υπάρχουν αρκετά πράγματα, μπορώ να σας πω ήδη τώρα. Τρία σημαντικά σημεία, δύο αρνητικά και ένα θετικό ως προς το Σύνταγμα της Ουγγαρίας. Επικρίσεις. Διατυπώσαμε στη γνωμοδότησή μας ήδη από ε, στο στάδιο της διαδικασίας έγκρισης του νέου συντάγματος. Αυτό που μας ανησυχούσε δηλαδή ήταν ότι το σχέδιο του συντάγματος ε, δημοσιεύτηκε στις 14 Μαρτίου, το δε σύνταγμα στο σύνολό του υιοθετήθηκε, εγκρίθηκε στις 18 Απριλίου. Δηλαδή για την συζήτηση ενός τόσο περίπλοκου και σημαντικού ε, νομοθετικού κειμένου μόνο πέντε εβδομάδες χρόνος διατέθηκαν και ίσως να μην αρκούσαν για το κοινοβούλιο, αλλά πάντως σίγουρα δεν αρκούσαν για τον δημόσιο διάλογο στην κοινωνία των πολιτών. Και αυτή ήταν η μία από τις ανησυχίες μας. Βέβαια, είχε προηγηθεί μία μακρά περίοδος συζητήσεων επί των αρχών μια γενικής, ενός γενικού διαλόγου για την ιδέα ενό νέου συντάγματο. Πάντως, η ουσιαστική συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο όταν έχει κατατεθεί ένα συγκεκριμένο κείμενο, πάνω στο οποίο μπορούν να τυπωθούν προτάσει και σχόλια. Δεύτερη ανησυχία ήταν αυτή σχετική με το σταγματικό δικαστήριο. Ήδη με το προηγούμενο σταγμα υπήρχε περιορισμός ε, των δικαιωμάτων του σταγματικού δικαστηρίου και τώρα πια αυτό δεν έχει τη δυνατότητα της πλήρους ε, του πλήρους ελέγχου, του σταγματικού ελέγχου ορισμένων κανόνων όπως των, κανόνων, των ε, νόμων περί εφαρμογής του, κανονι... του προϋπολογισμού ή ορισμένων που έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή μόνο σταγματικότητα συγκεκριμένων δικαιωμάτων μπορεί να επαληθεύσει το σταγματικό δικαστήριο. Έχει εξαιρεθεί, Φερρυπίνο, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, που είναι θεμελιώδες δικαίωμα και άρα ε, ανησυχούμε ότι δεν θα υπάρχει επαρκής προστασία της κυριότητας των δικαιωμάτων στην ιδιοκτησία εάν αποκλειστούν από το στοχματικό έλεγχο αυτά τα δικαιώματα. Θα σας υπενθυμίσω ότι έχει βρει τον τρόπο να αντιπαρέλθει αυτή την απαγόρευση στο στοχματικό δικαστήριο διότι ήδη έχει ακυρώσει ένα τέτοιο νόμο λόγω παραβίασης της αρχής ε, της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ένα άλλο ζήτημα αναδιοργανώνεται το δικαστήριο. Ήταν ε, η Ουγγαρία το μόνο κράτος που είχε τη λεγόμενη άκτιο ποπουλάρης, δηλαδή τη δυνατότητα για κάθε πολίτη να ζητήσει την αναθεώρηση για λόγους συνταγματικούς μιας, ε, ενός νομοθετήματος. Ε, αυτό τώρα αντικαθίσταται ως ε, διαδικασία από την ε, διαδικασία της ατομικής σταγματικής προσφυγής που υπάρχει στο γερμανικό δίκαιο και μπορεί ο καθένας να ζητήσει, ο κάθε να ζητήσει για λόγους παραβίαση των ατομικών του δικαιωμάτων ή των θεμελιωδών του δικαιωμάτων κάποιων σταγματικών αρχών τη σχετική ε, παρέμβαση του Σταγματικού Δικαστηρίου. Για την άλλη έκθεση, όπως σας είπα, δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες, αλλά κάποιες ιδέες μόνο που θα μας απασχολήσουν και θα ε, αποτελέσουν τη βάση της διατύπωσης αυτής της νομοδότησης. Για το προήμιο του συντάγματο αυτού, το οποίο είναι μακροσκελέστατο και έχει πολλέ ιστορικέ αναφορέ, έχουν εκφραστεί πολλέ ανησυχίε. Βέβαια, αυτό είναι χαρακτηριστικό σε ένα σύνταγμα κυρίω των νεαρών δημοκρατιών. Η ιδιαιτερότητα τη Ουγγαρία, δε είναι ότι στο σύνταγμα αυτό ένα άρθρο ρητά ορίζει ότι θα πρέπει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται υπό το φως του προημίου. Και πρέπει να επισημάνουμε τα εξή. Στο προήμιο υπάρχει ορισμός του έθνους, που ενδέχεται να ερμηνευθεί ως αποκλείον ορισμένες μειονότητες και δεύτερον, στο προήμιο αναφέρεται ότι έχει τεθεί εκτός ισχύω το Συντάγμα του 1949. Αυτό είναι πρόβλημα ω προ το εξή. Όχι γιατί δεν θέλει κανείς, γιατί θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τα κομμουνιστικά συντάγματα, αλλά γιατί έχει ορισμένε διατάξει που είναι ακόμη ενισχύ και άρα δεν είναι δυνατόν που θα έπρεπε μάλλον να μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί ή να τεθεί εκτός ισχύω καλύτερα ένα ε, σύνταγμα. Ένα άλλο ζήτημα που τίθεται είναι αυτό των Ούγγρων της Διασποράς και την ευθύνη για τις Ουγγρικές Αρχές να προσφέρουν προστασία στους Ούγγρους της Διασποράς. Αυτό το άρθρο μπορεί να θεωρηθεί ζήτημα κίνδυνος παρέμβαση στα εσωτερικά άλλων κρατών μελών. Τώρα, ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχουν συζητηθεί στο δημόσιο χώρο, στο δημόσιο διάλογο, Τώρα αναφέροντά τα δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι είτε τα επικρίνω είτε τα εγκρίνω. Απλώ να σα πω ότι είναι αντικείμενο συζήτηση. Ε, Καταρχά, το Σύνταγμα προβλέπει την προστασία του αγέννητου εμβρίου. Δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα για ισόβια κάθερξη χωρίς δυνατότητα ε, αποφυλάκησης, ε, συντόμευσης της ποινής ε, ή για λόγους καλής συμπεριφοράς. Δηλαδή μέχρι τέλους της ζωής ουσιαστική ε, ισόβια κάθεξη. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με σεξουαλικές ε, προτιμήσεις ή προσανατολισμό των ε, πολιτών, ότι δηλαδή αυτό το θέμα δεν έχει ενταχθεί στο άρθρο το σχετικό με την απαγόρευση των διακρίσεων, αλλά υπάρχουν άλλες αναφορές που θα μπορούσαν να καλύψουν την, σε σεξουαλικό προσανατολισμό. Η δε οικογένεια περιγράφεται ως ένωση μεταξύ ανδρός και γυναικός στο Σύνταγμα. σε άλλη κατηγορία τώρα του Συντάγματος, σε άλλο τμήμα, το, η δικαστική εξουσία. Στη δικαστική εξουσία σημειώνεται ότι είναι πολύ περιορισμένες οι λεπτομέρειες που αναφέρονται από το Σύνταγμα για την ε, λειτουργία, για τον τρόπο οργάνωσης δικαστικής εξουσίας. Δεν δίνει επαρκή περιγραφή του δικαστικού συστήματος. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόθεση για μια ευρύτατη και εκτεταμένη αναθεώρηση του δικαστικού συστήματος στην Ουγγαρία κάπου το φθινόπωρο και είναι πολλοί εκείνοι ε, στην Ουγγαρία που θεωρούν ότι χρειάζεται αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση του δικαστικού, ε, της, δικαστικής, της δικαιοσύνης. Απλώς είναι πολλά θέματα εκρεμεί ακόμη με αυτή τη νέα διατύπωση του συντάγματος και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η νέα μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Κρίσιμο σημείο πάντως είναι το έτος της ε, συνταξιοδότησης των δικαστών που από 70 μειώνεται στα 62 έτη ηλικίες, δηλαδή 300 από τους πλέον πεπειραμένους δικαστές, από τους ανώτατους δικαστές, θα υποχρεωθούν μέσα σε ένα χρόνο να εγκαταλείψουν την θέση τους, να βγουν στη σύνταξη, πράγμα το οποίο ε, υποθέτουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του δικαστικού συστήματος. σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές αρχές που είναι επίσης πολύ σημαντικές ε, τώρα, υπάρχει εν γέννη ένα σύστημα οργανικών θα λέγαμε νόμων, ε, κύριων νόμων, δηλαδή αυτών οι οποίοι πρέπει για να εγκριθούν να ε, έχουν την υποστήριξη των δύο τρίτων ε, των μελών του Κοινοβουλίου με ειδική πλειοψηφία. Και με το νέο σύνταγμα Υπάρχουν 56 αναφορές ή παραπομπές σε τέτοιου είδους οργανικούς νόμους. Δηλαδή θα υπάρξει τεράστιος αριθμός οργανικών νόμων που ουσιαστικά δεν υπάγονται πλέον στο δημόσιο διάλογο, στο, στην αναθεώρηση της δικαιοσύνη σε παραδείγματι. Ε, την έχει αναθέσει το νέο σύνταγμα την αναθεώρηση αυτή σε ε, τέτοιου είδους οργανικούς νόμους που όπως είπα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σε μια νέα πλειοψηφία ε, για τα θέματα τα σημαντικά να υπάρχει συζήτηση και να μην αρκεί μόνο μια υψηλή πλειοψηφία την οποία τώρα διαθέτει η κυβέρνηση για να εγκριθεί ένας τέτοιο νόμος. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για συζήτηση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, με την ε, σύνταξη, με τα διάφορα δικαιώματα. Ε, εκεί λοιπόν έχουμε πρόβλημα ως προς τους, οργανικούς αυτούς νόμους. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό του προϋπολογισμού, τον οποίο λαμβάνει κάποιος, ε, ε, κάποιο μεμονωμένο άτομο, ο πρόεδρος δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας με, με ένα συμβούλιο, το οποίο μπορεί να αποφασίσει αν υπάρχει πρόβλημα ως προς την τήρηση των κανόνων περί δημοσίου ελλείμματο και αν ασκήσει βέτο στο σχετικό προπολογισμό ή την εκτέλεσή του, δυνάμει τη ε, μη τήρηση των κανόνων περί δημοσίου ελλείμματο μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Και πάλι ερχόμαστε λέει, στο θέμα της δημοκρατίας και των, και ε, νομών που εγκρίνονται με δύο τρίτων πλειοψηφία. Επίση, υπάρχει μια προσέγγιση της τοπικής αυτοδιοίκησης πολύ κεντρική, άνωθεν επιβάλλονται οι κανόνες, δεν υπάρχει συμμετοχή της βάσης και νομίζω ότι το κείμενο το σχετικό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε τοποθέτηση, όπως είπα, συγκεκριμένη. Η γνωμοδότηση μας θα εγκριθεί 17 με 18 Ιουνίου. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι δεν έχει κλείσει η υπόθεση αυτή. Είναι πολλές και σημαντικές οι υποθέσεις που θα ε, υπαχθούν σε αυτούς τους οργανικούς νόμους που πρόκειται να υιοθετηθούν και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε όλοι να επαγρυπνούμε και να παρακολουθούμε τις διαδικασίες ε, έγκρισης αυτών των ε, οργανικών νόμων και να μην επαφεθούμε μόνο, να μην επαφεθούμε μόνο στην παρακολούθηση αυτής της συνταγματικής διαδικασία. Θα υπάρχει δουλειά και για μετά. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος για τους συντονιστές. Ως ήθιστε δίλεπτο ο καθένας διότι δεν είναι το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, μας μένει ένα για το ΕΛΚ. Η κυρία Γκάλλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο για αυτά που μας είπε, για την, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Βενετίας για, που αναφέρθηκε στο έργο αυτής της Επιτροπής. Επί σειρά ετών παρακολουθώ τις εργασίες της Επιτροπής αυτής. Αυτό που με ανησυχεί στη σημερινή συζήτηση είναι ότι δεν νομίζω ότι είναι της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να ασχολείται με το Ουγγρικό Σύνταγμα διότι εάν θέλουμε να συζητήσουμε οδήποτε στοιχείο ή λεπτομέρεια του συντάγματος του Ουγγρικού, αν δεν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε για οποιοδήποτε άλλο σύνταγμα χώρας της Ευρώπης. Κάποιες από τις επικρίσεις που ακούστηκαν ίσως να ισχύουν και για άλλα συντάγματα. Κάθε σύνταγμα Είναι θέμα κυριαρχίας συγκεκριμένης χώρας. Το επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος Μπαρόσο στις 5 Μαΐου στην Ολομέλεια. Είπε τότε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ασχολείται με εθνικά συντάγματα. Προφανώς είναι σημαντικό τα εθνικά συντάγματα να συνάδουν με διεθνείς υποχρεώσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με το Ουγγρικό Σύνταγμα. Δεν περιέχει διάταξη αντίθετη προς τις διεθνείς υποχρεώσεις. Ούτε προς τις υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που ανέφερε ο κύριος Μάρκατ είναι ζητήματα για τα οποία μόνο ερωτήσεις μπορώ να θέσω. η Επιτροπή της Βενετίας είπε σε απάντηση τριών τεθισών ερωτήσεων ότι δεν υπάρχει γενικός κανόνας σχετικά με τη διαθέτηση αυτών των ζητημάτων και πώς καλύπτονται αυτά από ευρωπαϊκά συντάγματα, όπως π.χ. ποια είναι η αρμοδιότητα του συνταγματικού δικαστηρίου. Και παραθέτω, συγκεκριμένες λεπτομέρειες αυτής της αναθεωρήσεως δεν μπορεί να συμπεριφθούν. Αν αυτό αληθεύει, δεν μπορούμε να μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα, αλλά δεν βλέπω γιατί ένα σύνταγμα είναι καλύτερο ή ανώτερο από κάποιο άλλο. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για άλλα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Παραδείγματο χάρη για το πώς αντιμετωπίζονται οι μειονότητες. Στην κεντρική Ευρώπη είναι μοναδικό το Σύνταγμα της Ουγγαρίας, διότι δηλώνει ότι οι εθνικοί Ούγγροι αποτελούν ένα κομμάτι του έθνους. Και ακόμα και τα συντάγματα της Σλοβακίας, της Μακεδονίας, λέει και της Ρουμανίας αναφέρουν, έχουν αναφορές σε μειονότητες. Νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα αλλά δεν νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση δικαιολογείται επ, αυτών, επ αυτής της βάσης. Αυτό το σημείο αναφέρθηκα. Δεν το τελευταίο σημείο στη μερίσια διάταξη, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε κρεμές σημείο της Βερονίκ Ματιούε. Περιοριστείτε λοιπόν παρακαλώ στις παρεμβάσεις σας. S&D, Φρασίκο Βαμπένοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την εκθέση. Ε, περιμέναμε κάτι πιο πλήρες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε. Σε ό,τι αφορά ε, στα όσα είπε η, η θέση των σοσιαλιστών και δημοκρατών δεν είναι εναντίον της δημοκρατίας της Ουγγαρίας ή εναντίον των πολιτών της χώρας, αλλά θα πρέπει να συζητάμε θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Ουγγαρία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν με άλλα κράτη-μέλη. Έτσι κάνουμε τώρα και με την κατάσταση της Ουγγαρίας. Ακούσαμε το πώς ε, έτυχε προετοιμασίας και υιοθετήθηκε το Σύνταγμα. Συμφωνούμε με τον Γραμματέα της Επιτροπής Βενετίας και θα θέλαμε όλα αυτά να καταγραφούν στην έκθεση της Επιτροπής. Ελπίζουμε ότι το πώς υιοθετήθηκε το Σύνταγμα θα αποτελέσει τμήμα της έκθεσής σας. Μας ανησυχούν ορισμένα ζητήματα. Το Σύνταγμα δεν περιλαμβάνει αρχές ε, διατάξεις για την προστασία των μειονοτήτων, για παράδειγμα ε, ε σε, για το... Ε, με βάση τις εξοβαλικές επιλογές των ατόμων. Ε, ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα λοιπόν δε, των ε, πολιτών δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα παρόλο ότι αφορά μια συγκεκριμένη μειονότητα. Δεύτερον σχόλιο. Το άρθρο Δέλτα, το οποίο αναφέρατε και το οποίο δεν ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο ε, και προβλέπει ε, ε εφαρμογή. Προβλέπει την υποστήριξη στην δημιουργία αυτόνομων περιοχών εκτός Ουγγαρίας κατά την, βασιζόμενο στην ε, συλλογική δράση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα διεθνή ε, κείμενα. Ευχαριστώ κυρία Ιντβέλτ. Μπορώ να είμαι σύντομη πρόεδρε. Ευχαριστώ τον γραμματέα για την παρουσίασή του. Συνηθίζουμε να εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένα, συγκεκριμένες πτυχές του συντάγματος, αλλά η ανησυχίες δεν πιστεύετε ότι αφορούν πιο πολύ την διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνονται αυτά τα στοιχεία του συντάγματος. Γιατί ξέρω ότι έχει πει η Ουγγρική κυβέρνηση, αν κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως υπάρχει σε κάποιο άλλο σύνταγμα, αλλά ο συνδυασμός τους είναι που μας δημιουργεί την ανησυχία. Δεύτερον, μας ανησυχεί η διαδικασία. Ε, η βεβαιασμένη αυτή διαδικασία με τις οποίες εγκρίθηκε το Σύνταγμα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας δικαστικής προσφυγής. Μετά, σε ό,τι αφορά τους, τις ε, κριτικές που απευθύνουμε, εμείς επικρίνουμε και τις δικές μας κυβερνήσεις, ακόμα και όταν το δικό μας κόμμα ήταν στην κυβέρνηση το επικρίναμε. Γιατί λοιπόν υπάρχει α, έκπληξη για το ότι συζητούμε το Ουγγρικό Σύνταγμα. Αν δεν συζητάμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, τι θα συζητάμε. Δηλαδή, γιατί συζητάμε όταν κάποιο κράτος μέλος παραβιάζει κανόνες όπως αυτών των κρατικών ή τους κανόνες ανταγωνισμού κλπ. Και δεν θα συζητάμε το, αυτό το σοβαρό ε, ζήτημα ή ξαφνικά η συζήτηση για αυτό το σύνταγμα γίνεται, ε, θεωρείται συζήτηση ε, επίθεση εναντίον τη Ουγγαρία. Χαίρομαι που κάθεσαι δίπλα μου γιατί μπορώ και σε κοιτάω εύκολα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να τα συζητάμε αυτά πολιτισμένα και να τα αντιμετωπίζουμε ως ε, συζήτηση που προστατεύει τη δημοκρατία στην Ευρώπη και όχι ως επίθεση εναντίον της Α ή της Β χώρας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, που δεν είναι. Ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε, ε, συζητήσεις αυτές να λαμβάνουν χώρα σε πιο αρμονική ε, ατμόσφαιρα, ε, πιο φιλική ατμόσφαιρα. Αυτό δεν κάνουμε άλλωστε και με τις υποψήφιες χώρες. Κοιτάμε τα συντάγματά τους, την ομοθεσία τους, συζητάμε ευαίσθητα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να είμαστε, την ίδια διαδικασία και με εμάς τους ίδιους. Ευχαριστώ κυρία Αργεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι εξελέγει με δημοκρατικό τρόπο η Ουγγρική κυβέρνηση. Όμως, για μία περίοδο τετραετή και όχι για πάντα εξελίγει για τετραετία. Και αυτή η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δείχνει ότι εργάζεται πολύ σκληρά και κινείται πολύ γρήγορα. Και φαίνεται σαν να βρήκε κάποια κολπάκια, ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι αν δεν είναι την επόμενη φορά το μεγαλύτερο κόμμα, ότι παρόλα αυτά θα εξακολουθεί να έχει κάποια εξουσία, διότι έλαβε τα μέτρα της. Κάποια απολύθηκαν από δικαστήρια ε, και μπορούν να υιοθετηθούν μόνο κάποιοι κανόνες μέσω πλειοψηφίας δύο τρίτων. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό όμως. Η δημοκρατία επιτρέπει να εγκρίνεις ή να απορρίψεις ε, νόμους κάθε ε, μερικά χρόνια και να γίνονται αλλαγές. Αυτό εμποδίζεται εδώ. Μπορείτε να μιλήσετε για διάκριση κατά των ομοφιλοφίλων ε, για το δικαίωμα της άμβλωσης για εθνοτικές μειονότητες, για το δικαστικό τομέα, τους δικαστές, για διάφορα θέματα, όμως στο κάτω-κάτω βλέπει κανείς ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να εξακολουθεί να κυβερνεί με μη δημοκρατικό τρόπο πέρα από την παρούσα θητεία της. Ας σκεφτούμε άλλες χώρες, όπως χώρες στην Αφρική, τον Μουμπάρακ ε, στην Αίγυπτο ή ηγέτες που εκτοπίστηκαν τώρα στην, ε, τους ηγέτες της Τινησίας. Τι να πούμε αυτές τις χώρες. Αυτά που λέγαμε αυτές τις χώρες πρέπει να μπορούμε να τα πούμε και για την Ουγγαρία. Έχω ένα ερώτημα για τους συναδέλφους και για την Επιτροπή της Βενετίας. Τι περιθώριο έχουμε πέρα από αυτό το ηθικό ε, θέμα να μιλήσουμε κατά της απομάκρυνσης από την δημοκρατία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Επιτροπή της Βενετίας τα Ταβάρες. Καμιά φορά τέτοιος ευρύς ορισμός της κυριαρχίας και αυστηρή εφαρμογή της επικουρικότητας χρησιμοποιείται. Όπως αυτό που είπε ο συνάδελφος Κίγκεργάλ, αν κολλήσουμε σε αυτά τα πρότυπα, αποδυναμώνουμε εντελώ τι διατάξει τη συνθήκη περί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αν τα συντάγματα είναι τέτοιο εργαλείο κυριαρχία που είναι ε, στεγανά και δεν μπορούν να είναι αντικείμενο κριτικής απ' έξω, τότε μπαίνουμε στον κόσμο της συνταγματικής σχετικότητας που οδηγεί σε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω συντάγματος. Και δεν μπορούμε να το επικρίνουμε αυτό. Διότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το πορτογαλικό σύνταγμα με το Γκρικού και να πούμε ότι το πορτογαλικό είναι καλύτερο. Ε, είναι σχετικισμός αυτός, είναι σχετικότητα συνταγματική. Εμείς υιοθετήσαμε στην Πορτογαλία καινούριο σύνταγμα μετά από δικτατορία. Μετά το τέλος της δικτατορίας μάλλον. Και είχα καλωσορίσει συζητήσεις επί του δικού μας συντάγματος. Και το πώς υιοθετούνται αυτά τα συντάγματα. Ο κανόνας των δύο τρίτων είναι σημαντικό κανόνας. Πρέπει να προσέξουμε όμως το πνεύμα που κρύβεται πίσω από τον κανόνα. Δηλαδή πρέπει να εξασφαλίζει συνένεση και διαρκείας μάλιστα χρονικής. Τι συμβαίνει όταν ένα κόμμα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων. Μπορείς να μπλοκάρεις για περίοδο ε, χρονική κάποια βασικά κείμενα. Άρα έχουμε σε δύο πτυχές. Ρήτρα μη διάκρισης δεν αρκεί. Δεν αρκεί να λέει κανείς ότι αφαιρούμε τη σεξουαλική προτίμηση από τη διάκριση, αλλά ε, δεν υπάρχει καμία άλλη διάκριση. Δηλαδή εξαρτάται από την ερμηνεία ενός δικαστηρίου η, η προστασία από διάκριση παρά να καθορίζεται σαφώς από το Σύνταγμα. Από τους οργανικούς νόμους διέπονται πολλά. Άρα πρέπει να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με αυτούς τους οργανικούς νόμους, διότι πολλά που συγκρούονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα πλαισιώνονται από τους οργανικούς νόμους. Άρα πρέπει να συζητήσουμε και τους οργανικούς νόμους όπως θα ε, εφαρμόζονται στην ε, Ουγγαρία. Πρόεδρος, ακολουθούμε συγκεκριμένη γραμμή. Αυτή θα ακούσουμε πρώτα όλου αυτού που είναι στον κατάλογο που βάλουν σε ερωτήσει πριν να ακούσουμε την απάντηση. Αυτή είναι η γραμμή που ακολουθούμε. Λοιπόν, ο κύριο Μπουσετήλ είναι επόμενο. Το ΕΛΚ ε, διστάζει πάντα ε, σε να διεξάγουν τέτοιου συζητήσει γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι αρμοδιότητά μα να συζητάμε ένα σύνταγμα ε, ενό συγκεκριμένου κράτου μέλου. Παρ' όλα αυτά η πλειοψηφία διαφώνησε με την άποψή μα. Οι συνάδελφοι είπαν ότι έχουμε αρμοδιότητα να εξετάζουμε την διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ σήμερα, αλλά έχοντας ακούσει την παρουσίαση του γραμματέα της Επιτροπής Βενετίας, ε, ε, είδαμε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δεν υπάρχει θέμα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ό,τι κατάλαβα. Το πολύ πολύ να υπάρχει κριτική ότι η διαδικασία διήρκεσε μόνο πέντε εβδομάδε, αλλά δεν βλέπω παράβαση ανθρωπίνων, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτό, ούτε και ελέγχθη κάτι τέτοιο. Το δεύτερο παράπονο ε, ακόμα δεν έχει ε, εξεταστεί πλήρως ε, από την Επιτροπή. Θα δημοσιευθεί το πόρισμα τον Ιούνιο. Οπότε το ελάχιστο που θα πρέπει να κάνουμε θα ήταν να περιμένουμε τη δεύτερη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βενετίας και μετά να συζητήσουμε το θέμα. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα πράγματα σχολιάστηκαν από το γραμματέα. Για παράδειγμα, προστασία της ζωής που δεν έχει γεννηθεί, των παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί αν εξετάσουμε αυτό το σύνταγμα για αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να εξετάσουμε και το ελληνικό σύνταγμα για το ίδιο ζήτημα. Γιατί δεν συζητάμε το ελληνικό και κανεί δεν το ζητάει. Επίση γίνεται αναφορά για την ε, διάκριση με βάση των σεξουαλικών επιλογών, ότι αυτή η, ε, η μη διάκριση δεν συμπεριλαμβάνεται. Ας δούμε και άλλα συντάγματα, τα οποία δεν έχουν τέτοιου είδους αναφορές. Αυτό από μόνο του αποτελεί διάκριση επί τη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού. Μετά, ε, γάμος μεταξύ άνδρα, ανδρών και γυναικών μόνο. Και πάλι να εξετάσουμε πολλά, τέτοια, πολλά συντάγματα που έχουν παρόμοιες διατάξεις. Είναι πώς. Η Σοφή Ιντβέλτ ε, έθεσε το δάχτυλο επί των τύπων των Ήλων. Ε, είπε ότι αν δεν συζητούμε τις αξίες μα, περί είναι η Ευρώπη. Αυτό ακριβώ σοφή. Οι δικέ μας αξίες είναι διαφορετικές από τις δικές σου και θα πρέπει να δεχτείς ότι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικέ χώρε έχουν διαφορετικέ αξίε. και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα, ε, μία βασική ε, οριζόντια αρχή. Ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα και όσο πιο σύντομα αρχίζουμε, αρχίσουμε να σεβόμαστε τις διαφορές ακόμα και στις αξίες μας τόσο πιο γρήγορα θα μάθουμε να συζούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κ. Μωράης. Um, Θα αλλάξω λίγο τα όσα είχα να πω ε, για να τα προσαρμόσω. Καταρχήν, ε, να ξεκαθαρίσω, να ξεκαθαρίσω το εξή. Από όταν έγινα μέλο, έχουμε συζητήσει επανειλημμένω το Ιρλανδικό Σύνταγμα, τι επιπτώσει του. Έχουμε συζητήσει ορισμένα πολύ ευαίσθητα θέματα που προκύπτουν από το Ιρλανδικό Σύνταγμα για τη σεξουαλικότητα, για τα γέννητα ε, παιδιά κλπ. Συνεπώς, δεν συζητούμε τις, ε, τα διαφορετικά νομοθετικά κείμενα απλώς διαφορετικών χωρών. Αυτό που ζητάμε από την Επιτροπή της Βενετίας είναι να μας συγκρίνει και να μας αναλύσει το κατά πόσον η διαδικασία του συντάγματος ήταν ορθή, το κατά πόσον ε, είναι θεμητό οργανικοί νόμοι να ρυθμίζουν πολλά ευαίσθητα θέματα. Ε, αναφερθήκατε, ε, κύριε Γραμματέα, για πολλή ώρα στους οργανικούς νόμους, ακριβώς επειδή είναι πολλά τα ζητήματα που καλύπτουν. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Ε, ο διορισμός των δικαστών. Αν καθορίζεται ένα όριο συνταξιοδότησης ηλικιακό όριο, θα ήθελα να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμητό να αναλύσουμε ένα σύστημα μέσω του οποίου χρειάζονται, ε, χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων για την ψήφιση των οργανικών νόμων και να το συγκρίνουμε με άλλα, με άλλα συντάγματα, κάτι το οποίο κάνετε. Και είναι θεμητό να αναλύουμε το κατά πόσον αυτό ε, έρχεται σε αντίθεση ή είναι συμβατό με τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει των συμβάσεων που έχουν υπογράψει. Συνεπώ, δεν συζητούμε τις διάφορες χώρες, τα διάφορα νομοθετικά κείμενα. Συζητάμε το κατά πόσον ένα σύνταγμα ε, είναι συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή όχι. Και σίγουρα δεν μπορούμε να ε, ξετάσουμε το θέμα του προπολογισμού ε, ή άλλων ζητημάτων προκύπτουν από το Σύνταγμα, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούμε να τα συζητάμε. Επίση, ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά του οργανικού νόμου και την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων. Υπάρχει άλλο Σύνταγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυτή τη διαδικασία. Thank Κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βλέπω να έρχεται εδώ στην Επιτροπή μας η Επιτροπή της Βενετίας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που είχατε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε μας και διαβάζω εδώ το φυλάδιο και είναι πολύ εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο ε, γίνεστε παγκόσμια εμβέλεια και προσελκύεται και μέλη εκτός Ευρώπης, προφανώς λόγω της ποιότητας των εργασιών σας. Αυτό είναι πόλος έλξης. Είναι πολύτιμο αυτό. Θα ήθελα να δω μια ανάλυση της Επιτροπής της Βενετίας όσον αφορά το Σύνταγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, που δεν είναι γραπτό, είναι πασίγνωστο. Ίσως κάνατε, αν ψάξω την ιστοσελίδα, να βρω κάποια μελέτη σας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η δουλειά που κάνετε είναι πολύ αυστηρή ε, και αμερόληπτη ε, πνευματικά και δημιουργικά. Δεν μεροληπτείτε, αλλιώς δεν θα προσελκύετε και μέλη εκτός Ευρώπης. Και η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Συμβουλίου της Ευρώπης, η συνεργασία που αυξάνεται είναι ευπρόσδεκτη. Συναντηθήκαμε και με μέλη του δικαστηρίου, τα μέλη της ΛΥΜΠΕ. και με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, στο δικαστήριο αυτό τα πράγματα είναι ακόμα πιο σημαντικά. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Μάλλον Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Σάιμον είπε κάποια πράγματα σωστά. Υπάρχει όριο αμφισβητούμενο μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνταγματικών προτύπων και πολιτισμικών αξιών. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ε, υπογράψει τη συνθήκη, είναι όλα μέλη της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Συμβάσης τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και εκεί συμπεριλαμβάνεται σαν θέμα η μη διάκριση. Άρα είναι σαφές τι έχουμε υπογράψει νομικώς πώς και ποια είναι η ακριβής, η ακριβής εφαρμογή είναι θέμα ερμηνείας των όσων υπογράψαμε. Ήθελα να τα πω ξεκάθαρα όλα αυτά. Ευχαριστώ η κυρία Μποτσκούχα, έχει το λόγο. Μάλιστα. Ε, πράγματι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη στην ε, ποικιλία, στην, στην... αλλά πρέπει να βρούμε τα σημεία που μας ενώνουν παρά εκείνα που μας χωρίζουν. Ένα από αυτά τα σημεία είναι ότι όλοι έχουμε βασιστεί στα θεμελιώδη δικαιώματα, δημοκρατία, ή στα δικαιώματα για τους πολίτες. Αυτές είναι οι κοινέ μας αξίες που μας ενώνουν. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Όλοι υπερασπιζόμαστε αυτές τις ιδέες. Και νομίζω ότι αυτή είναι και αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Εμείς πολεμάμε για τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Έχω συγκεκριμένο ερώτημα προς την Επιτροπή της Βενετίας. Μια εποχή που συζητούμε τα ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα σεξουαλικής προτίμησης, προσανατολισμού. Κάτι που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς είναι δυνατόν να συζητούμε εδώ άλλους λόγους, άλλες βάσεις, άλλα αίτια τα οποία μπορούν να εισάγουν ε, κάποιες ανισότητες. Ευχαριστώ ως Μπρόγκς. Η Ουγγρική κυβέρνηση αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ εθνικότητας και υπηκότητας και ηθαγένειας μάλλον, που είναι συγκεκριμένα στη Δύση. Τα πρώτα μέσω οικογενειακής ε, σχέσεως αποκτούν, τα δεύτερα μέσω γεννήσεως ή μέσω ε, νομικής πράξης. Λοιπόν, οι, οι πρόγονοι των Ούγγρων που έχουν μεταναστεύσει ε, ήταν θύματα αλλαγή συνόρων ε, μετά τη συνθήκη του 1920. Δεν έφυγαν εθελοντικά. Είναι φυσικό να θέλει να τους φροντίσει η Ουγγρική κυβέρνηση. Θα να προστατεύσει τους ε, ομοεθνείς τους, κυρίως ε, διότι καμιά φορά είναι αντικείμενα καταπιεστικής ε, νομοθεσίας αυτή. Ο κύριος Γκόνς, η κυρία Γκόνς μάλλον, τα τελευταία λόγια. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Κοιτάξτε, ε, άλλη μια πτυχή θέλω να τονίσω που αφορά το ογκρικό Σύνταγμα. Αναφέρατε, κύριε Γραμματέα της Επιτροπής τη Βενετία, σημαντικές στοιχείες. Αυτή την ξεχάσατε. Είχε τέσσερι θέσει διαμεσολαβητή η Ουγγαρία μέχρι τώρα. Γενικό διαμεσολαβητή, υπεύθυνο μετά για την μειονότητα, για τι μειονότητε, ένα για τι μελλοντικέ γενιέ και ένα διαμεσολαβητή για την προστασία των δεδομένων. Πολύ ισχυρή θέση αυτή. Σημαντικότατη εποχές αλλαγών. Ήταν σημαντικότατο θέμα, το θέμα της των δεδομένων, το, το πιο σημαντικό επί σειρά ετών. Τώρα αντικαθίστανται από διαφορετικό σύστημα δημοσιολαβητών. Έχουμε γενικό δημοσιολαβητή με δύο βοηθούς, που είναι, ένας είναι για τις μειονότητες και για μελλοντικέ γενιές και δεν ο άλλος δεν υπάρχει διαμεσολαβητής για την προστασία των δεδομένων. είναι ανεξάρτητη η θέση του διαμεσολαβητή. Είναι υπόλογο μόνο στο κοινοβούλιο. Κάποια αρχή αντικαθιστά τους άλλους διαμεσολαβητές. Εμείς ασχολούμαστε με την προστασία των δεδομένων. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Με αυτή την αλλαγή τι γίνεται τώρα είναι το ερώτημα. Πώ διευθετείτε το θέμα τη προστασία των δεδομένων μετά την αλλαγή που έγινε με του σε αυτό είναι το ερώτημα. Δίνω το λόγο στον κύριο Μάρκετ, λέει ο πρόεδρο, για να συνοψίσει. Όσο πιο σύντομα γίνεται, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ε, ε ήταν συνάντηση ενημέρωση τώρα. Δεν αποφασίζουμε τίποτα. Στο κάτω-κάτω περί ενημερώσεω πρόκειται. Μπορώ πολύ εύκολα να είμαι σύντομο, καταρχά, διότι εκπροσωπώ το Συμβούλιο της Ευρώπης και ετοιμάζουμε μια γνωμοδότηση για την κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν έχουμε έρθει για να παρέμβουμε στη δική σας συζήτηση. Ήρθαμε γιατί μας καλέσατε και εσείς θα αποφασίσετε εάν θέλετε να χειριστεί το θέμα αυτό ή όχι. Άρα δεν μπορώ να σας σχολιάσω. Δεύτερον, δεν έχουμε ακόμη υιοθετήσει την ε, γνωμοδότησή μας και ως εκ δεν μπορώ να επισέλθω στα διάφορα ζητήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα καταλήξουμε ή θα διατυπώσουμε τα συμπεράσματά μας. Οφείλουμε να περιμένουμε μέχρι ότου ετοιμαστεί η δική μας γνωμοδότηση. Ένα ερώτημα νομίζω ήταν είναι συγκεκριμένο του κυρίου Μωράης. Με συγχωρείτε, δεν λυγιμονήσα την ερώτηση όμως. Α, ναι, για τους ε, οργανικούς νόμους. Το θυμηθήκατε. Ναι, όντως, δεν υπάρχει άλλη χώρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει τόσο ευρύ φάσμα ε, οργανικών νόμων. Από την άλλη υπήρχαν ε, και στο παρελθόν στην παράδοση την νομική της Ουγγαρίας αυτή η οργανική νόμη και άρα ερχόμαστε στο θέμα που θέτει η κυρία Ινερτφέλντ ή ο κύριος Τάβαρες ότι είναι πολλά τα ευρωπαϊκά συντάγματα τα οποία στηρίζονται στην στο αξίωμα ότι αρκούν τα δύο τρίτα της πλειοψηφία για να παρουσιάσουν μια εικόνα συνένεσης ε, προκειμένου να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσει. Τώρα, για λόγου που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει μόνη σε αυτά δύο τρίτα τη πλειοψηφία. Κάποιε διασφαλιστικέ δικλείδε μπορεί να λειτουργούν, κάποιε όχι. Δεν θέλουμε να παρεμποδίσουμε τη διαδικασία του συντάγματος. Ίσως θα ήταν από πλευρά εκείνων οι οποίοι έχουν την ε, πλειοψηφία αυτών δύο τρίτων το καλύτερο να ήταν να απόσχουν από την άσκηση της εξουσίας τους με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τίποτα τέτοιο δεν έχουμε δει ακόμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μάρκερτ, την Επιτροπή της Βενετίας, αυτού του συμβουλευτικού οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παραμένουμε, διατηρούμε ανοιχτή τη γραμμή δεν έχει κλείσει το θέμα αυτό και δεν έχουμε τη συζήτηση αυτή για να, για να αποφασίσουμε να κρίνουμε κάτι η ενημέρωση αυτή παραμένει ανοιχτή. Έχουμε ακόμα δύο-τρία λεπτά, αν μου επιτρέπετε. Να το αναβάλουμε, λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Κύριε Ματσιέ. Και αν δεν υπάρχει τίποτε άλλο στο διάφορο, Διακόπτεται η συνεδρίαση. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη. Χαίρετε.